C'est trois fois. Bonjour. La réunion... Καλημέρα σας. Ο πρόεδρος μας είναι στη Ουάσιγκτον. Δεν υπάρχουν αντιπρόεδροι, άρα θα πρέπει να αρκεστείτε στους πρεσβύτερους σήμερα. Πρώτο θέμα, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Όσον αφορά την ημερήσια, θα ήθελα να σας πω ότι εξαιτίας ε, της ηλεκτρικής βλάβης της Δευτέρας και επειδή ακριβώς δεν μπορέσαμε να εγκρίνουμε δύο εκθέσεις, Γκίγολτ ε, και Κάζα, θα ψηφιστούν σήμερα από τις 12 παρατέταρτο. Υπάρχουν σχόλια σε σχέση με την ημερήσια διάταξη. Φαίνεται πως όχι, άρα εγκρίνεται. Δεύτερον, ανακοινώσεις της Πρόεδρου. Θα πρέπει να σας πω καταρχήν ότι ο τελευταίος τριμερής διάλογος για την οικονομική διακυβέρνηση έγινε χτες και η πρόεδρος, ο πρόεδρος ε, θα μιλήσει για τις συμφωνίες και θα γίνει μια επαναδιαβούλευση, επαναδιαπραγμάτευση τη Δευτέρα 26 2011. Άρα θα γίνει νέα διαβούλευση μαζί σας. Ως προς τις ε, συνεδριάσεις μας για το 2012 έχετε το χρονοδιάγραμμα όπου υπάρχει ένα λάθος που εγκρίθηκε στις, ε, όπως ξέρετε στις 11 Ιουλίου για τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012 η συνεδρίαση θα γίνει το απόγευμα και όχι το πρωί όπως αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα και θα σας αποσταλεί ένα διορθωτικό. Τρίτη ανακοίνωση. Θα γίνει μία ανοιχτή συνεδρίαση των συντονιστών με τον Επίτροπο Σεμέτα στις 6 Οκτωβρίου από τις 9.30 στις 11. Και ο Επίτροπος θα μας ενημερώσει για την πρόταση της Επιτροπής για τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Γιατί η πρόταση αυτή θα δημοσιευτεί μία μέρα πριν. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και θα δούμε τι χειραγωγήσεις έχει κάνει η Επιτροπή επί του θέματος σε σχέση με αυτό το φόρο ως προς τον ε, τριμερή διάλογο για τις ανοιχτές ε, πωλήσει, short selling, έγινε μια συνεδρίαση για τις ανοιχτές ε, πωλήσει στις 20 Σεπτεμβρίου. Πήλθε πρόοδος, όμως παρά τις συζητήσεις δεν έγινε καμία, δεν υπήρχε καμία συμφωνία σε σχέση με τις ανοιχτές πωλήσει. Συμφωνήθηκε ότι τα τρία θεσμικά όργανα θα συνέλθουν για να επιτύχουν έναν συμβασμό. Το ΕΛΚ ζήτησε opt-out ενώ το Συμβούλιο θα επιθυμούσε το αντίθετο. Άρα οι διαπραγματεύσεις θα διαρκέσουν τρεις μήνες. Ο επόμενος τριμερής διάλογος θα γίνει τον Οκτώβριο και θα οριστεί η επακριβή ημερομηνία. Αυτά ως προς τις ανακοινώσεις ε, της Προέδρου. Ε, υπάρχουν σχόλια, εάν όχι, θα φτάσουμε στο τρίτο θέμα που είναι η δημόσια ακρόαση για τη συλλογική προσφυγή σε σχέση με τα αντιτράστ. Εδώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον ε, Επίτροπο Αλμούνια που είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής υπεύθυνος για τον ανταγωνισμό. Εκείνος έχει περισσότερες αρμοδιότητες κρίνω και θα μας κάνει μία εισήγηση. Μετά θα, θα ακούσουμε τον κύριο Κρέστορ Χότς, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Φιλίπ Ντεγκούχτ και ε, τον κύριο Κόενς, τέλος. Ah, λοιπόν, πρώτα θα ακούσουμε τον Επίτροπο. Ε, Κύριε Σβάμπ, θέλετε να κάνετε μία εισαγωγή. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εντάξει. Θα ακούσουμε τον Επίτροπο. Ε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτά τα εισαγωγικά σας σχόλια. Κυρίες και κύριοι, Κύριε Βουλευτές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να ανταλλάξω με απόψεις μεταξύ μας όσον αφορά τη συλλογική προσφυγή. Με μεγάλη χαρά βλέπω ότι το Κοινοβούλιο δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό ε, και υποβάλλει προτάσεις ε, έτσι ώστε και εμείς με τη σειρά μας να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον προβληματισμό των ε, καταναλωτών πρόκειται ε, για ένα θέμα το οποίο πρέπει να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ε, Ο κύριος Επίτροπο μιλάει, λέει η πρόεδρο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Continue. Ε, Έλεγα λοιπόν ότι έχω την εντύπωση ότι οι συζητήσεις καμιά φορά για το θέμα αυτό ξεχνούν ότι πρέπει να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Η ενίσχυση του νόμου που διέπει τον ανταγωνισμό ε, έχει δύο σκέλη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει και την Κομισιόν και τις Εθνικές Αρχές ε, οι οποίες εφαρμόζουν τα ίδια άρθρα των συνθήκων ε, και έχουν ένα πολύ καλό και υψηλό επίπεδο συνεργασίας χάρη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού. Επίσης έχουμε και το τους, ε, την ιδιωτική δυνατότητα η οποία προσφέρεται από την εθνική νομοθεσία. Θέλω να πω ότι στην Ευρώπη δεν ε, υπάρχει ίδια δυνατότητα προσφυγής ε, σε περίπτωση που παραβιαστεί ο κανονισμός αντιτράστ σε οποιοδήποτε όμως μέρος της Ευρώπη, Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν ζει κανείς ε, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα και να προσφεύγει σε υπόθεση αντιτράστα αλλά και να ε, έχει αποζημίωση. Θα πρέπει επομένως να υπάρξει μεγαλύτερη σχέση ανάμεσα την δημόσια δυνατότητα παρέμβασης και την ιδιωτική. Ε, και η συλλογική προσφυγή είναι μια πάρα πολύ καλή γέφυρα ανάμεσα στα δύο. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις απέναντί μας και θα σας πω ποιες είναι και πώς μπορούμε να τις ε, αντιμετωπίσουμε. Ε, οποιαδήποτε προσφυγή μπορεί να ξεκινήσει πριν ή και αφού ξεκινήσει μια διαδικασία επιπαραβάση από τις αρμόδιες αρχές αυτό είναι απαραίτητο γιατί θέλουμε να παραμείνουμε ε, στην γραμμή των προγραμμάτων μας τα οποία κύριο στόχο έχουν την καταπολέμηση των καρτέλ. Βεβαίως ε, οι περισσότερες διαδικασίες ε, λαμβάνουν χώρα αφού ξεκινήσει μια εθνική αρχή την αντίστοιχη δράση και βεβαίως μπορούν να υπάρξουν προσφυγές σε μερικές περιπτώσεις πριν οι δημόσιες αρχές αρχίσουν από μόνες τους να λαμβάνουν, ε, ε, να λαμβάνουν μέτρα. Ε, σε μερικές χώρες μπορούν να ξεκινήσουν ε, ε, γρήγορα οι διαδικασίες ενώ σε άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία επί πριν φτάσει στο δικαστήριο ε, η προσφυγή αυτή. Με τον τρόπο αυτό καθυστερούν πολύ οι διαδικασίες σε όλα τα εθνικά δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύω ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλες ομάδες οι οποίες να ε, γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίζουν τα θέματα των ε, προσφυγών ε, θα πρέπει όπως έλεγα και στην αρχή να υπάρξει και συνέργεια ανάμεσα στις δημόσιες συλλογικές διαδικασίες και τις ιδιωτικές διαδικασίες. Εμείς ε, έχουμε προχωρήσει ε, στο, μέσω του συστήματος, του ευρωπαϊκού συστήματος επίλυσης ε, διαμαχών, έχουμε προχωρήσει σε συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες δυσκολεύουν την δυνατότητα καταχρηστικής θέσης. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει και η απαραίτητη γνώση των δικηγόρων όσον αφορά τις καταχρηστικές ε, διαφωνίες ε, και την δυνατότητα εξοδικαστικής επίλυσης των διαφωνιών. Πιστεύουμε ότι η καλή γνώση και οι σωστές δράσεις είναι αυτές οι οποίες θα διασφαλίσουν ε, την ορθή χρήση του συστήματος ποια είναι τα επόμενα βήματα. Όπως γνωρίζετε, η Κομισιόν προτίθεται να εγκρίνει μία ανακοίνωση όσον αφορά τη συλλογική προσφυγή μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Ε, και συνεργάζομαι και με την συνάδελφο Ρέντιν και τον Επιτροπό Νταλή όσον αφορά τα ε, θέματα αυτά. Ε, γιατί βεβαίως και το περιβάλλον και η προστασία των καταναλωτών είναι σκέλη της Επιτροπής ανταγωνισμού θα πρέπει να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε ε, σε όλες τις ανάγκες ε, και τις απαιτήσεις ε, και των ιδιωτικών και των συλλογικών προσφυγών και από αυτού πρέπει να πω ότι και στις δύο περιπτώσεις η δράση μας θα πρέπει να είναι πολύ πιο έντονη ε, στην ε, έκθεση ανταγωνισμού που εγκρίνατε πέρυσι ε, καλή για συγκεκριμένες νέες δράσεις όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού και όσον αφορά και την συλλογική προσφυγή. Οπωσδήποτε θα εφαρμοστούν αυτές οι νέες αρχές στην συλλογική προσφυγή αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει και ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκη εξειδίκευση ε, και λεπτομερής ε, κατάλογος δεσμευτικών και μη δεσμευτικών κειμένων περί ανταγωνισμού. Επ' αυτού τελειώνω και ε, περιμένω να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρόεδρος, θα δώσω τώρα τον λόγο στον επόμενο ομιλητή. Για πέντε λεπτά θα έχει το λόγο. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Uh, I should also... Θα για να σας κάνω ευτυχής, να σας πω ότι είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Έρασμος στην Ολλανδία. Θα πρέπει να δούμε πώς να αποφύγουμε τις συλλογικές προσφυγές στην Ευρώπη. Και εάν μιλήσουμε για ένα ξεχωριστό σύστημα συλλογικών προσφυγών, είναι σαφές ότι εκεί όπου υπάρχει ζημία θα πρέπει να υπάρχει και αποκατάσταση της ζημίας και αποκατάσταση της αγοράς που θα πρέπει να προτρέχει των αναγκών της αγοράς. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για την επιβολή του νόμου. Η συλλογική προσφυγή αφορά ένα ιδιωτικό ένδικο μέσο. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς εφαρμόζονται αυτά τα ιδιωτικά μέσα και αν πρόκειται για τον δημόσιο ή το ιδιωτικό τομέα. Το νομικό σύστημα των ΙΠΑ είναι υπέρ της ιδιωτικής εφαρμογής και οι Αμερικανοί δεν θέλουν να εφαρμόζεται το δίκαιο από ομοσπονδιακές αρχές οι οποίες είναι ε, στο έλεος του, της εκτελεστικής εξουσίας. Από την άλλη πλευρά τα δικά μας συστήματα, το ευρωπαϊκό σύστημα, είναι είτε της ιδιωτικής και της δημόσιας εφαρμογής του δικαίου. Γι' αυτό οι αμερικανικές τεχνικές όπως οι συλλογικές πρόσφυγες ήταν ένα ένδικο μέσο που δεν προβλεπόταν στην Ευρώπη. Όμως τα ευρωπαϊκά δίκαια πολλές φορές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν πολύπλοκα και συλλογικά θέματα. Στην, ε, στη ΣΥΠΑ ε, δημιουργείται και υπάρχει αυτός ο μηχανισμός με βάση μια διαδικασία opt-out. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι υπέρ των συλλογικών προσφυγών και τις έχουν εφαρμόσει τα τελευταία δέκα χρόνια. Αλλά δεν χρησιμοποιούνται τακτικά διότι το χρηματοοικονομικό σκέλος δεν είναι δελεαστικό έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί από τους συνήγορους. Υπάρχει ένα ιδιαίτερα υψηλό κόστος που για μας φαίνεται κάτι το καταχρηστικό. Η θεωρία των ΙΠΑ αφορά μέτρα αναχέτησης σε σχέση με εφαρμογή μέτρων ex Σε αντίθεση με αυτό, πολλοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί πέρα από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού έχουν μία επιτροπή έχουν μία εφαρμοστική, ένα εφαρμοστικό δίκαιο, ας το πούμε, το οποίο δεν βασίζεται σε μέτρα αναχέτησης. Κατά την άποψή μου, η θεωρία και μόνη της αναχέτησης είναι πιο δαπανηρή και δεν μπορούμε να βασιστούμε αποκλειστικά σε αυτήν, διότι πρόκειται για μία προσέγγιση ex post και υπάρχουν πολλές κυρώσεις και μεγάλο κόστος για την ανείχνευση των ε, παραπτωμάτων και παρατυπιών. Εάν θέλει κανείς να ενθαρρύνει τις ιδιωτικές συλλογικές προσφυγές, θα πρέπει να άρει τα προσκόμματα προς τον ενάγοντα και να δώσει κίνητρα και στους ενάγοντες και στους συνήγορους έτσι ώστε να μπορέσουν να επιλύσουν με αυτό το μέσον τις διαφορές. Αυτό ακριβώς κάνει το σύστημα των ΙΠΑ. Αυτά τα προσκόμματα είναι οικονομικής υφής. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερο κόστος προς τον ενάγοντα και υψηλά τέλη ή ε, υψηλές αμοιβέ. Και επίσης μέσα στα πλαίσια των αποζημιώσεων δεν θα πρέπει να έχουμε μία μακροχρόνια διαδικασία στα πλαίσια της επίλυσης της διαφοράς. Εάν εισαγάγουμε τους ανωτέρω μοχλούς θα μπορούσαμε να ε, αποθαρρύνουμε το πλαίσιο αυτό χρήσης. Ε, δεν υπάρχουν ε, άλλες ρήτρες διασφάλισης. Θα πρέπει να παίξουμε με αυτούς τους μοχλούς. Οι μοχλοί αυτοί βρίσκονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί θεωρούν ότι αυτοί οι μοχλοί δεν υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό είναι μεγάλο λάθος. Υπάρχουν σαφείς στάσεις σε πολλά κράτη-μέλη. Δεν, υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει βοήθεια προς τον ενάγοντα. Και εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε χαμηλό κόστος μεταφόρας και να έχουμε και χρηματοδότηση από τρίτα μέρη ή ε, μεσολαβητές, ενδιάμεσους. Εμείς προσπαθούμε να εισαγάγουμε αυτή την νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης υπάρχουν και άλλοι μοχλοί όπως η μεσολαβητες ενδιαμεσους εμεις προσπαθουμε να εισαγαγουμε της υπόθεσης, η πιστοποίηση από το δικαστήριο, opt-in ή opt-out, προγενέστερες ανακοινώσεις, έγκριση από το Δικαστήριο των Αμοιβών των Δικηγόρων και ε, απόφαση επί της συνέχειας που θα δοθεί σε μία διαφορά. Όμως, κανένας από αυτούς τους μοχνου, μοχλούς δεν μπορεί να διαβαθμιστεί είτε μεμονωμένα είτε σωρευτικά από τεχνικής ή οικονομικής πλευράς. Ένα σύστημα δεν μπορεί να δώσει ε, αρκετές διασφαλίσεις γιατί θα έχετε ή πολύ λίγα ή πολλά στην εφαρμογή μέσα στα πλαίσια της θεωρίας αναχέτησης και αυτό εξαρτάται από τις αξιώσεις που υπάρχουν στους διάφορους τομείς. Δηλαδή, αν προβάλλετε περισσότερους μοχλούς, ίσως, ίσως διαγκωθεί και η διαφορά. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς έχουν τα εσωτερικά ένδικα μέσα των κρατών μελών η επιβολή του δικαίου ανταγωνισμού αφορά οποιοδήποτε ένα δίκαιο όπως όλα τα άλλα. Σε αυτή την περίπτωση η μοχλή είναι ακριβώς η ίδια. Σε αυτή την ιδιαίτερα ατυχή περίπτωση θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι εναλλακτικές που διαθέτουμε. Υπάρχουν μερικές. Οι συλλογικές προσφυγές, η συλλογική προσφύγη είναι μια πεπαλαιωμένη τεχνική και υπάρχουν τώρα πιο σύγχρονα συστήματα. Μία εναλλακτική προσέγγιση, η οποία ήδη χρησιμοποιείται σε ορισμένα κράτη-μέλη, αλλά όχι ακόμα ευρέως στο τομέα του ανταγωνισμού, αφορά την ιδιωτική εφαρμογή, που δεν είναι και το μόνο μέσο που διαθέτουμε. Φαίνεται από την έρευνα ότι οι ρυθμιστές μπορούν να προβάλλουν αποζημιώσεις σε συλλογικές προσφυγές και μπορούν να το κάνουν τάχιστα και χωρίς υψηλές δαπάνες όταν έχουν τα κατάλληλα μέσα. Πολλές φορές όμως τα ε, συμβαλόμενα, μάλλον οι αντίδικοι, μπορούν να βοηθηθούν από τον ε, διαμεσολαβητή, ο οποίος έχει την κατάλληλη πραγματογνωμοσύνη. Εάν οι ρυθμιστές έχουν δυνατότητες επιβολής των μέτρων, όπως ισχύει στην περίπτωση της Δανίας με την Telecom και τα συστήματα RDR είναι πολύ πιο γρήγορα για την αποζημίωση. Εάν χρειάζονται νέες διαδικασίες σε έναν μεμονωμένο ε, τομέα μέσα στα πλαίσια συγκεκριμένων μηχανισμών πολλές φορές δεν βοηθά τους πρωτογενείς μηχανισμούς αποζημιώσεων. Δεν θα πρέπει λοιπόν οι συνήγοροι να ζητούν αυτό τον μηχανισμό και θα πρέπει να προβάλλεται μόνο αν δεν υπάρχει η τεχνική RDA Ορισμένα ε, δικαστήρια το προβλέπουν σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Χρειάζεται αποζημίωση η οποία θα πρέπει να προβάλλεται γρήγορα και χωρίς υψηλές δαπάνες. Δυστυχώς όμως υπάρχουν πεπαλαιωμένες τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται. Και αυτό αφορά και τα μέτρα επιβολής που προβάλλονται μέσα από τις αποφάσεις των συλλογικών προσφύγων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φιλίπ Ντεμπούκ έχει το λόγο που είναι γενικός διευθυντής της Business Europe, ο οποίος έχει τέσσερα λεπτά στη διάθεσή του. Έχετε το λόγο. Μην χάνετε χρόνο ψάχνοντας το μικρόφωνο, λέει η Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ε πρόεδρε, Αντιπρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης ε, που έχει την ευκαιρία να εκφραστεί και η Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Κοινότητα. Όπως γνωρίζετε ανέκαθαν ήμασταν υποστηριχτές και της οικονομίας, της αγοράς άρα και των πολιτικών ανταγωνισμού. Ήμασταν ε, θερμοί υποστηρικτές και της εσωτερικής αγοράς αλλά και των καλών σχέσεων με την καταναλωτική κοινότητα η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι εκ των όνου κάνευ για να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους. Και ε, το θέμα που μας απασχολεί σήμερα θα συνεισφέρει και πρέπει να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση αυτή και το στόχο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, άρχισε μια διαβούλευση και έκανε πολλές ερωτήσεις. Βέβαια δεν έχω χρόνο, γι' αυτό θα επικεντρωθώ σε δύο μόνο. Πρώτον, οι συλλογικέ αγωγές θα πρέπει να είναι ένα μέσο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Εμείς έχουμε την άποψη και μάλιστα την έντονη άποψη ότι η επιβολή του νόμου θα πρέπει να παραμείνει αυστηρά στα χέρια των κρατικών αρχών. Ειδικό του ρόλο είναι και είναι σε καλύτερη θέση να εγγυώνται ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Γι' αυτό η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να σταματήσει να ε, να αποφύγει μάλλον να διολυστήσει προς την ιδιωτική επιβολή του νόμου. Υπάρχουν αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού και είναι δική τους δουλειά. Το να περάσουμε τώρα σε ιδιωτική ε, εφαρμογή θα ε, σημαίνει μεγαλύτερη δικαστική ε, επέμβαση πολλά κράτη αυτόν τον καιρό προσπαθούν να μειώσουν τους διακανονισμούς γιατί έχουν έξοδο για την κοινωνία. Υπάρχουν και ε, καταχρήσεις που ε, έχουν ως στόχο μόνο το οικονομικό συμφέρον των μεσολαβητών. Θα πρέπει να αποφύγουμε συλλογικές ε, δικαστικές διαδικασίες που είναι πάρα πολύ χρονοβόρες και πάρα πολύ βαριές διαδικασίες και τελικά είναι μικρή αποζημίωση για τα θύματα. Θα ήθελα και πάλι να τονίσω, με επιτρέπετε, ότι Είναι βεβαίως σημαντικό να αποζημιώνονται εκείνοι ε, που πέφτουν θύματα κάποιων που παραβιάζουν τον νόμο. Σωστό είναι αυτό. Ωστόσο δεν επιλέγουμε εμείς ε, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον τρόπο και το μέσο των συλλογικών προσφυγών ή αγωγών. Το ε, θέμα τώρα η πρόθεση δεν είναι να αρχίσει ένα τέτοιο σύστημα στην Ευρώπη με όλα τα στοιχεία όμως που έχουμε δει υπάρχουν ή θα μπορούσαν να ε, ε, υπάρξουν. Αν γίνει μια τέτοια συλλογική προσφυγή στη δικαιοσύνη για ένα σύστημα στην Ευρώπη εγκατασταθεί, δεν θα μπορέσουμε να φύγουμε τα περίφημα τοξικά, όπω λέγονται, στοιχεία που συνδέονται με τι συλλογικέ αγωγέ. Η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να το επιβάλλει αυτό το σύστημα, αλλά μπορεί να επιβάλλει και όλα τα ειχέγγια και τι ασφαλιστικέ δικλίδες που ανέφερε προηγουμένω και ο Καθηγήτη ε, για τα έξοδα τα δικαστικά, για τι διαδικασίε αποκάλυψη. Όλα αυτά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και άλλα, όχι μόνο αυτά. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και άλλες λύσεις που έχουν ήδη ακουστεί. Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ στο ADR που είναι η εναλλακτική ε, μορφή επίλυσης ε, των διαφορών. Είναι πιο ρεαλιστικό, πιο αποτελεσματικό και ε, σήμερα το πρωί μια πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Ρέντινγκ. Τελειώνω. Αυτό το σύστημα EDR μπορεί να σημαίνει ταχεία και αποτελεσματική και φτηνή αποζημίωση των καταναλωτών σε μια εσωτερική αγορά. γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις αυτόν τον καιρό για το θέμα και στο Κοινοβούλιο και εκτός και ε, το υποστηρίζουν πολύ ενδιαφερόμενοι και οι καταναλωτές. Γι' αυτό αξίζει να ε, διερευνήσουμε τα ωφέλη από το σύστημα αυτό και ε, σε περιπτώσεις ε, ανταγωνισμού. Επιτρέψτε μου να τελειώσω λέγοντας ότι η Business Europe βεβαίω είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα εξώδικο όμως μέσο που ε, θα σημαίνει ταχεία και αποτελεσματική αποζημίωση χωρίς να μπούμε σε θέματα διενέξεων και διακανονισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Διευθυντά, λέει η Πρόεδρος. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μονή Γκέρνς από την Ευρωπαϊκή ε, Οργάνωση Καταναλωτών. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε και μια γυναίκα, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ του mainstreaming. Βέβαια, μπορείτε να ε, θεωρήσετε ότι η γυναίκα ε, αξίζει όσο τρεις άντρες, έτσι, ε, σε ό,τι αφορά την ισορροπία του φίλου. Εγώ δεν είμαι εδώ ως γυναίκα, ως εκπρόσωπος των καταναλωτών είμαι και θα ήθελα να σας δώσω και τη φωνή εκείνων που πέφτουν θύματα χρήσεων ανταγωνισμού. Ε, και για μένα βεβαίως είναι μεγάλη υπόθεση και δυσκολία να σας δώσω τις απόψεις μας σε τέσσερα λεπτά. Και έχουμε κάποια καρτούν εδώ, κάποιες γελιογραφίες και ε, ε, στοιχεία, αλλά θα τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας. Η ε, συλλογική δράση και οι συλλογικές αγωγές ε, σε θέματα ανταγωνισμού και κατάχρησης μπορεί κάποιος να τα θεωρεί πάρα πολύ θεωρητικά και εγκεφαλικά, αλλά συμβαίνει στην καθημερινή ζωή. Να σας δώσω παραδείγματα. Πριν από λίγους μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε ένα πρόστιμο 300.000 ευρώ 300 εκατομμύρια, συγγνώμη, για μια εταιρεία που παράγει απορριπαντικά. Γιατί ε, κανόνιζαν τις τιμές, έκαναν συνεννοήσεις και όλοι έχετε χάσει τουλάχιστον λίγα ευρώ το χρόνο επειδή υπήρχαν συνεννοήσεις στα θέματα των τιμών των απορριπαντικών. Βεβαίως δεν θα πάει κανείς στο δικαστήριο χέφρον για λίγα ευρώ, αλλά τελικά πρόκειται για εκατομμύρια ε, παράνομα κέρδη και αυτά θα πρέπει να... Ε, πληρωθούν ως πρόστιμο. Το πρόστιμο επευλήθη, αλλά τα θύματα δεν αποζημιώθηκαν. Αυτό είναι το θέμα λοιπόν των συλλογικών αγωγών προσφυγών. Και το δικό μας μήνυμα είναι πολύ απλό. Όταν κάποιος είναι θύμα ενός ε, τέτοιου φαινομένου, κατάχρησης ε, της ε, σπόζουσας θέσης ας πούμε, θα πρέπει να αποζημιώνεται και θα πρέπει οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να το ζητούν. Βεβαίω μπορεί να υπάρχει ένα φιλικό διακανονισμό ω πρώτο βήμα με τι εταιρείε και πρέπει να πούμε ότι μετά την απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πήγαμε στις αρμόδιες εταιρείε και αυτοί αρνήθηκαν να κάνουν φιλικό διακανονισμό με τους καταναλωτές γιατί είπαν ότι δεν τους έβλαψαν. Για ποιο λόγο. Εκεί ε, το χάσαμε αυτό. Συμφωνούμε ότι το ADR είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο η εναλλακτική δηλαδή μορφή επίλυσης των φορών αλλά σε συλλογικές ε, δράσεις και προσφυγές δεν είναι ίσως το καλύτερο. Ε, η δημόσια επιβολή είναι το καλύτερο, αλλά ξέρετε τι πόρους έχουν τα κράτη. Είναι γνωστά αυτά και δεν μπορούν οι καταναλωτέ να εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών για το αν θα τους αποζημιώσουν. Αυτό λοιπόν. Οι συνολικές ε, δράσεις, οι συλλογικές ε, προσφυγές και αγωγές είναι ένα εργαλείο, αλλά υπάρχουν και άλλα συμπληρωματικά. Επίσης θα ήθελα να μιλήσω για αυτό το σύνδρομο των ε, Αμερικανικών ε, συλλογικών προσφυγών. Πολλοί μύθοι κυκλοφορούν στην Ευρώπη για το τι συμβαίνει στη ΣΥΠΑ. Εμείς έχουμε πολύ συχνά επαφές και με συναδέλφους εκεί και με τις κρατικές αρχές, αλλά και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ε, προχωρήσει ε, και σε άλλες ρυθμίσεις γιατί υπάρχουν και άλλα φαινόμενα όπως είναι οι εκβιαστικοί διακανονισμοί ε, και τέτοια φαινόμενα. Θα πρέπει στα κράτη-μέλη να είναι δεσμευτική νομοθεσία για να μπορούν να αποζημιώνονται συλλογικά οι καταναλωτές. Δηλαδή, οι οργανώσεις καταναλωτών να μπορούν συλλογικά να προσφεύγουν, πώς να το πω, Το δικαστήριο να αποφασίζει αν είναι περίπτωση opt-in ή opt-out, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις το opt-in δεν επιτρέπεται, δεν γίνεται. Να, ας πούμε για μερικά ευρώ, ε, είδατε αυτό που σας είπα για τα απορριπαντικά, δεν θα πάει κανείς να ε, ε, κάνει αγωγή στην εταιρεία για λίγα ευρώ. Ε, θα πρέπει επίσης σε θέματα τραστ ε, και καταπολέμησής τους να έχουν οι καταναλωτές και εκπρόσωποι τους καλύτερη ενημέρωση, πρόσβαση στα έγγραφα και χρηματοδότηση των μέσων αυτών. Και τέλος θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σωστό και συνεπές να έχουμε συλλογικές ε, ρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά υπάρχουν ε, ε, διάφοροι κλάδοι, προστασία των καταναλωτών, προστασία του περιβάλλοντος, ανταγωνισμός. Θα ήταν φιάλτης σε όλους αυτούς τους τομείς να έχουμε μια εγκάρσια, μια οριζόντια ρυθμίση. Τελειώνω, Πρόεδρε. Κοινέ αρχές λοιπόν με κλαδική νομοθεσία ζητούμε και όχι ένα τέτοιο εγκάρσιο σύστημα ε, συλλογικών προσφυγών για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε λοιπόν τι είχαν να μας πούν οι εμπειρογνώμονες. Όλα ήταν ενδιαφέροντα και σαφή. Θα ζητήσω πρώτα απ' όλα από τον εισηγητή, τον κύριο Σβάμπ, ε, Ανδρέα, θέλει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους ειδικού και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τα ενδιαφέροντα που μας είπαν. Νομίζω ότι στο Κοινοβούλιο συμφωνούμε όλο και περισσότερο ότι στην Ευρώπη θα πρέπει να αναπτύξουμε κοινέ αρχέ για τέτοιε συλλογικέ μορφέ διεκδίκηση. Ε, των δικαιωμάτων σε κάποια κράτη υπάρχει και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κρίστοφερ Χότς γιατί σήμερα τα συστήματα που ήδη υπάρχουν στα κράτη-μέλη συλλογικών προσφυγών γιατί έχουν μείνει χωρίς αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό και χωρίς επιτυχία. Ακούμε επιχειρήματα που λένε ότι όλα αυτά δεν είναι τόσο ξένα προς το κοινοτικό δίκαιο, αλλά δεν έχουν καμιά τεράστια επιτυχία. Πού οφείλεται αυτό. Δεύτερον, αυτές οι κοινέ αρχές που υποτίθεται ότι θα είναι σε ένα οριζόντιο μέσο δεν θα πρέπει να επικαλύπτονται και ευχαριστώ πολύ τον Αντιπρόεδρο κύριο Αλμούνια. Τα ειδικά θέματα που αφορούν το ευρωπαϊκό ε, δίκαιο ανταγωνισμού που διέπεται από την αρχή του public enforcement, δηλαδή της επιβολής από ε, τις δημόσιες κρατικές αρχές. Και επίση τα έγγραφα θα πρέπει να παραμένουν απόρριτα, αλλιώ ε, ποτέ κανένα δεν θα παραδεχτεί ότι στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Ξέρω ότι ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να διατηρήσουμε κάποια στοιχεία. Κύριε Αλμού, γιατί θα κάνετε εσείς. Γιατί ακούσαμε την κυρία Γκογιένς ε, να εκφράζει επικρίσεις για τις εγκάσεις, οριζόντιες ρυθμίσεις. Πώς θα εξασφαλίσετε τις ιδιαιτερότητε του δικαίου ανταγωνισμού. Και ένα τελευταίο που για μας όλους είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό τον καιρό. Στο θέμα των συλλογικών αγωγών ή προσφυγών είναι δύσκολο να έχουμε ενιαία θέση γιατί πλήττονται σκληρά οι εταιρείε από την κρίση και προσπαθούμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελαφρύνουμε τις επιχειρήσεις αντί να τις επιφαρύνουμε περισσότερο. Γι' αυτό θα πρέπει να επιλέξουμε ε, μια συνετή προσέγγιση και χαίρομαι που πρότεινε ο κύριος ε, Αλμούνια, κάτι που είχα προτείνει και εγώ στην γνωμοδότησή μου για την Επιτροπή αυτή. Τελικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχει ε, όφελος ο καταναλωτής αλλά και πολύ χαμηλό κόστος. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ντεμπίκ και την κυρία Γκόγιανς, έχετε ακούσει ε, στα κράτη-μέλη τι συμβαίνει σαν αυτό που μας είπατε με τα πορυπαντικά που οι καταναλωτές έχουν ο καθένας μικρή βλάβη, μικρή ζημία αλλά δεν έχουν κρατήσει τις αποδείξεις, ας πούμε, από πού αγόρασαν το απορριπαντικό για να πούνε πόσο το πλήρωσαν. Αυτό δεν θα πρέπει να ε, είναι προς όφελος του κράτους τελικά τα έσοδα από τα πρόστιμα, γιατί πού θα βρει τον κάθε καταναλωτή να τον πληρώσει. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Edith Λεπέλς, άλλοι θέλουν το λόγο. εντίτ και μετά ε, να απαντήσουν ε, οι εμπειρογνώμονε μας. Ευχαριστώ. Καταρχήν, ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχήν που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση γιατί μιλάμε για ένα άκρος ενδιαφέρον και σημαντικό θέμα η οικονομολόγος θα ήθελα να έχω μία άκρωση προσέγγιση επί του θέματος γιατί μιλάμε για καθαρά τομεακές, τομεακή προσέγγιση που ίσως είναι δυνατή στην Ουγγαρία. 400.000 οικογένειες έχουν πληγεί από το σύστημα υποθηκών και πολλοί ε, είχαν υποστεί ζημίες ως απότοκο αυτής της κατάστασης. Οι οικογένειες σκέφτηκαν ότι όταν ε, υποθηκεύσουν σε ξένο νόμισμα αυτό θα ήταν ε, ένα μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά οι καταναλωτές δεν είχαν τις σωστές πληροφορίες από τις τράπεζες εγκαίρως. Θα μπορούσα λοιπόν να πω ότι παραπλανήθηκαν οι καταναλωτές. Στη συνέχεια οι τράπεζες ε, συνέχισαν μόνο μερός να αλλάζουν τις συμβάσεις και όλο το κόστος αυτών των αλλαγών το υπομίστηκαν οι καταναλωτές οι ίδιοι, δηλαδή οι δανειολήπτες. Εδώ μιλάμε για επανόρθωση, για μέτρα επανόρθωσης μέσω συλλογικών προσφυγών. Θα ήταν δυνατόν να προβάλλουμε αυτή αυτά τα μέτρα σε μια τέτοια περίπτωση, δηλαδή συλλογική προσφυγή σε μια τέτοια περίπτωση. Ο κύριος Φεγιό έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας σε αυτό το συλλογικό μάθημα, σε αυτή τη μήνυα ακρόαση θα ήθελα και εγώ να ε, υποβάλω μία ερώτηση. Θα ήθελα να αναφερθώ στην Πορτογαλία, στη χώρα μου που γνωρίζω καλύτερα, όπου υπάρχει ένα ένδικο μέσο παρόμοιο με αυτό που λέτε, πρόκειται για τη λεγόμενη λαϊκή προσφυγή και μέχρι τούδε υπήρξαν δυσκολίες εφαρμογής καθώς και βασικές ελλείψεις στο σύστημα. Καταρχήν υπάρχουν προβλήματα αναγνώρισης, αναγνώρισης των ίδιων των εναγωμένων και είναι πολύ δύσκολο να οριστούν και οι ζημίες ποσοτικά και ποιοτικά. Καθώς και το ποιος έχει υποστεί βλάβη και πώς επακριβώς. Επίσης, τα ίδια τα δικαστήρια αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες για την επίλυση αυτών των διαφορών. Και με αυτές τις συλλογικέ προσφυγές α, βλέπουμε ότι υπάρχει μία δυσλειτουργία των εθνικών δικαστηρίων. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς μπορούμε να άρουμε αυτά τα προσκόμματα και τις δυσλειτουργίες δηλαδή κατά πόσο μπορεί να επιληθεί διαφορετικά μία διαφορά μέσω διαιτησίας, μέσω διαμεσολάβησης και ούτω καθεξής έτσι ώστε να μην ε, δημιουργήσουμε μία κατάσταση μόνιμης ρήξης και μόνιμων διαφορών. Πρόκειται για διαδικασίες που δεν θα πρέπει να είναι τόσο δαπανηρές. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω ότι σε έναν άλλο τομέα, σε θέματα φορολογικών διαφορών στη χώρα μου, για να πληθούν αυτές οι διαφορές χρειάζονται 10 χρόνια. Τώρα εφαρμόζεται ένα νέο πρόγραμμα το οποίο ορίζει ότι η διαιτησία θα πρέπει να εκτελεστεί, εκτελεστεί στα πλαίσια των φορολογικών διαφορών πιο γρήγορα, τουλάχιστον σε σχέση με τα 10 χρόνια που προβλέπονταν αρχικά. Euh, Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ράπτη έχει δει στο λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ είμαι φιλοξενούμενη εδώ, δεν εργάζομαι στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων που διοργανώνει την ακρόαση. Εργάζομαι στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς ε, η οποία θα έχει μία γνωμοδότηση για αυτό το θέμα των συλλογικών προσφυγών. Ε, βλέπω, αισθάνομαι ότι υπάρχει μία διάθεση να πυροβολήσουμε τις συλλογικές προσφυγές ε, δεν αισθάνθηκα καλά όταν άκουσα τον κύριο καθηγητή να χαρακτηρίζει πεπαλαιωμένο εργαλείο, παλιό εργαλείο, τις συλλογικές προσφυγές. Ε, νομίζω ότι κάθε εργαλείο έχει τη χρησιμότητά του ανάλογα με τον τρόπο και με το πώς χρησιμοποιείται το ADR είναι μια, ένα νέο εργαλείο, ένα μοντέρνο εργαλείο, για να χρησιμοποιήσω αντίστοιχη ανάλογη ε, ορολογία με τον κύριο καθηγητή, ε, το οποίο κατά τη γνώμη μου μπορεί να συνδυαστεί με επιτυχία με τις συλλογικέ προσφυγές. Εκτιμώ ότι το ADR μπορεί να είναι ένα πρώτο βήμα προσπάθειας για επίλυση διαφορών αλλά η συλλογική προσφυγή έχω την αίσθηση ότι πρέπει να υπάρχει διότι στην ευρώπη δεν υπάρχουν μόνο επιχειρήσεις μεγάλες υπάρχουν και οι καταναλωτές και υπάρχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εκεί ακριβώς θα ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο αλμούνια ο οποίος καταλαβαίνω ότι ε, το κύριο θέμα του είναι ο ανταγωνισμός και εγώ έχω στο μυαλό μου τον ανταγωνισμό πώς μπορούμε να συνδυάσουμε και τα δύο μέσα από μια οριζόντια προσέγγιση στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λεσμίκη είναι ο τελευταίος που ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που καθυστέρησα και ίσως να είμαι και λίγο προκατηλημένος άλλωστε γιατί είμαι υπέρ της συλλογικής προσφυγής εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί ξέρετε είναι κάτι το οποίο ε, ε επί σειρά ετών δεν ήθελε καμία πλευρά. Ε, η Business Europe ε, λέει και φαντάζομαι ότι και οι προηγούμενοι ομιλητές το ίδιο είχαν πει ε, ο, αναφέρεστε στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Ε, κατά την άποψή μου δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια ολοκλήρωση εάν δεν έχουμε δυνατότητα προσφυγής. Και αναρωτιέμαι γιατί φοβάστε τόσο πολύ τον κόσμο, τον απλό πολίτη, τον απλό πολίτη. Υπάρχουν πάρα πολύ κακά παραδείγματα στις ε, Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά υπάρχουν όμως και μερικές μερικά εξαιρετικά παραδείγματα, μερικές εξαιρετικές περιπτώσεις. Μπορεί να πει κανείς, εντάξει αυτό δεν μπορεί να συμβεί στην Ευρώπη, αλλά πιστεύω ότι τουλάχιστον τη δυνατότητα πρέπει να την έχουμε. Γιατί διαφορετικά δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ η ενιαία αγορά. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα δώσω το λόγο τώρα στους ε, εμπειρογνώμονες και όπως ο κύριος ε, Φιλίπ Ντεμπίκ πρέπει να φύγει, θα δώσω πρώτο τον λόγο σε αυτόν, σαν εκπρόσωπο της Business Europe και μετά θα δώσω το λόγο αμέσως στον Επίτροπο Αλμούνια. παρακαλώ, σας ετέθησαν ερωτήματα, αν μπορείτε να απαντήσετε. Ε, βέβαια όταν θα απαντήσει ο Επίτροπος εγώ θα έχω φύγει, αλλά τι να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής ε, για την δυνατότητα που μας έδωσε να ανταλλάξουμε απόψεις. Ε, ο Αντρέας Βάμπα βεβαίως έθιξε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα όσον αφορά ε, το θέμα της μικρής αποζημίωσης για πολύ κόσμο και αυτό είναι σημείο, στοιχείο κλειδί όταν μιλάμε για ανταγωνισμό. Μας απασχολεί, μας απασχολεί το θέμα αυτό και όσον αφορά τη συλλογική ε, προσφυγή Γι' αυτό λοιπόν ε, βλέπουμε και από κοντά τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε ε, τις ε, περιπτώσεις στρέβλους ανταγωνισμού και αντιτράστ λοιπά. Γιατί οι αποζημιώσεις όντως μερικές φορές είναι πολύ λίγα χρήματα για πολύ κόσμο. Ε, δεν ξέρω ε, τις λεπτομέρειες της δικιά σου περίπτωσης ε, Μονίκα, αλλά φαντάζομαι ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να κάνουν τέτοιες προσφυγές και αυτό θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ κακό για όλους. Δεύτερον, όσον αφορά τις τράπεζες και από όσο ξέρω ήδη υπάρχουν συλλογικές δράσεις ε, κατά των ε, τραπεζών, κυρίως ε, από τη στιγμή που το 2007-2008 ξεκίνησε η κρίση βεβαίως αυτές οι προσφυγές γίνονται βάσει των εθνικών νομοθεσιών και είναι γεγονός ότι κρατούν σε μάκρος οι διαδικασίες αλλά πάντως υπάρχει δυνατότητα προσφυγής για την Πορτογαλία, ναι, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα προς αποφυγήν, δηλαδή πώς δεν πρέπει να προχωρήσουμε. Ε, πρόσφατα σε ε, αντίστοιχη ακρόαση του Κοινοβουλίου ε, μια παρόμοια ε, άποψη εξεφράστη και από την ίδια την Πρόεδρο της Επιτροπής Εφαρμογής των Δικαστικών Αποφάσεων και της Πορτογαλίας και βεβαίως όπως είπα και προηγουμένως είναι γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει μεγάλη τοξική επίδραση τέτοιων προσφυγών. Η συλλογική προσφυγή είναι πεπαλαιωμένο. Δεν λέω ακριβώς αυτό. Λέμε ότι ενδεχομένως θα έπρεπε σαν σημείο εκκίνησης να μην διαλέξουμε τη συλλογική προσφυγή αλλά την εναλλακτική επίλυση διαφορών, το ADR. Γιατί βεβαίως ο θυγόμενος καταναλωτής θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αποζημιωθεί. Ε, για τον επόμενο ομιλητή ε, βεβαίως έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να προσφύγουν και δεν φοβόμαστε ε, τη δυνατότητα που θα έχει να προσφύγει ο μεμονωμένος πολίτης αλλά φοβόμαστε τις επιπτώσεις των πολλαπλών αγωγών και την στρέβλωση που ενδεχομένως θα προκύψει στην αγορά. Ε, εμείς κάναμε κάποιες ε, προτάσεις ε, και ακριβώς είχαμε ζητήσει να γίνει ενδελεχέστερη ανάλυση ακριβώς γιατί οι τοξικές επιπτώσεις μπορεί να είναι πολύ μεγάλες και γι' αυτό ακριβώς είπαμε ότι θα πρέπει σαν βάση να θεωρήσουμε καλύτερα την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Εν πάση περιπτώσει όμως η επιχειρηματική κοινότητα σαφέστατα είναι υπέρ των διαδικασιών αυτών ε, και οπωσδήποτε αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να φτάνουν σε κάποια, σε κάποια επίλυση. Ευχαριστώ. Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα αγγλικά. Θα αρχίσω απαντώντας την ερώτηση που μου έγινε απευθείας από τον κύριο Σφαπ Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του δικαίου ανταγωνισμού στην Ευρώπη ή πώς συνδέουμε την ε, επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού από το κράτος με τις αποζημιώσεις ε, σε περίπτωση παραβίασης στα θύματα. Πώς αυτά συνάδουν. Τα είπα στην αρχική μου τοποθέτηση. Η αποζημίωση και η αποκατάσταση μπορεί να γίνει, όπως και γίνεται άλλωστε σε πολλά κράτη-μέλη με διάφορους τρόπους, μέσω μεμονωμένων προσφυγών, ατομικών, εταιρείε που πηγαίνουν στα δικαστήρια γιατί ε, ζητούν αποζημίωση από άλλες εταιρείε που έχουν ε, οργανωθεί σε καρτέλ ή ε, παραβιάζουν το δίκαιο ανταγωνισμού και αυτό αποβαίνει εις βάρος κάποιων εταιριών, τις ανάγουν. Σε κάποιες περιπτώσεις Αυτές οι μεμονωμένες λοιπόν ατομικές δράσεις που βεβαίως είναι δαπανηρές για τον ενάγοντα μπορούν να γίνουν μόνο από εταιρείε. Είναι πάρα πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις όπου ένας πολίτης, ένα πρόσωπο έχει την οικονομική δυνατότητα και ρισκάρει να απευθυνθεί στο δικαστήριο για να αποσμειωθεί. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις αλλά δεν είναι ο κανόνας. Μεγάλες εταιρείε όμως έχουν ε, το δικαίωμα και μπορούν να το ε, ασκήσουν κιόλα. Τώρα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έπεσαν θύμα ενός καρτέλ ή πολίτες πάλι που έπεσαν θύματα ε, καρτέλ κατά 99% για να μην πω 99,9% δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους για να προσφεύγουν ατομικά. Γι' αυτό είναι αυτό το ερώτημα. Μπορούν να οργανωθούν συλλογικές δράσεις, συλλογικές αγωγές για να αποζημιώνονται αυτές οι περιπτώσεις. Όταν αποφασίζουμε για ένα πρόστιμο, ας πούμε, έχει διαπιστωθεί η παραβίαση, ο στόχος της επιβολής προστίμου όμως δεν είναι η αποζημίωση των θυμάτων. Ο στόχος μας όταν επιβάλλουμε ένα πρόστιμο είναι να αποτρέψουμε εκείνους που παραβιάζουν ε, την νομοθεσία να το επαναλάβουν και εκείνους που θα μπουν στον πειρασμό να τους αντιγράψουν. Η αποζημίωση δεν είναι στα χέρια μας όταν επιβάλλουμε πρόστιμα. Δύο λοιπόν είναι τα διαφορετικά την εδώ. Η εθνική νομοθεσία στα κράτη-μέλη μπορεί να διαφέρει στους τρόπους και στα μέσα που επιτρέπουν. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είπε ο καθηγητής Χότζες, υπάρχει ή υπήρξε μια εξέλιξη που μπορεί να θεωρηθεί ότι προσεγγίζει το σύστημα που ισχύει ε, την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά γνωρίζουμε, τουλάχιστον στην υπηρετική Ευρώπη, ότι το νομικό μας σύστημα δεν ταιριάζει με τέτοια συστήματα και τέτοιες διαδικασίες όπως αυτές που ε, ισχύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε. Αφενός να βρούμε κάποιες αρχές για ενός είδους συλλογική δράση και προσφυγή και στον τομέα του ανταγωνισμού για να προσπαθήσουμε να θεσπίσουμε κοινέ αρχές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως Μία από τις αρχές αυτές θα πρέπει να είναι σαφής δέσμευση ότι θα αποφεύγονται κάθε είδους καταχρήσεις που γνωρίζουμε ότι υπήρξαν στο παρελθόν ή εξακολουθούν να υπάρχουν στο σύστημα των ΗΠΑ. Εγώ είμαι πολύ πιο αισιόδοξο από τον κύριο Ντεμπούκ. Ο κύριος Ντεμπούκ είναι προσιλωμένος στην παλιά πρόταση Μα δεν εργαζόμαστε στην παλιά πρόταση. Εμείς κάναμε δημόσια διαβούλευση και μάλιστα ευρύτατη και εργαζόμαστε στην εκπόνηση κοινών αρχών για μια ανακοίνωση. Και η συνάδελφος Βιβιάν Ρέντινγκ που είχε αντίστοιχη ακρόαση ε, σε ε, ε, επιτροπή πριν το καλοκαίρι το ίδιο είπε. Συνεργαζόμαστε πολύ επιτροπή, κυρία Ρέντινγκ, ο κύριο Ντάλι και ο υποφαινόμενο για να καταθέσουμε αυτέ τι κοινέ αρχέ μετά από μια ευρύτατη δημόσια διαβούλευση. Οι περισσότεροι από του ενδιαφερόμενου που ρωτήσαμε, με εξαίρεση ε, του επιχειρηματίε που εκπροσωπούνται από την Business Europe, οι περισσότεροι λοιπόν ενδιαφερόμενοι συμφώνησαν ότι υπάρχει ανάγκη να βρεθούν κάποιε κοινέ αρχέ. Ακόμα δε, δεν έχουμε αποφασίσει ποιο θα είναι το επόμενο βήμα για τις συλλογικέ προσφυγές. Θα λάβουμε εσωτερική απόφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα για αυτές τις αρχές. Θα τις δημοσιεύσουμε σε μια ανακοίνωση και στα πλαίσια αυτού του διαλόγου που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα τονίσουμε τις ιδέες μας. Αν αρκούν αυτοί οι κανόνες για να τους λάβουν υπόψη τα κράτη-μέλη και να τους ενσωματώσουν στην εκάστοτε νομοθεσία τους ή όπως είπε ένα συνάδελφό σας στην έκθεσή του, ο κύριος Λένε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, ε, αν χρειάζεται ένα νομικό οριζόντιο μέσο κτλ. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα ως εκεί. Κοινέ αρχές όμως χρειάζονται. Το επόμενο θέμα, ιδιαιτερότητες του ανταγωνισμού για ε, αποζημίωση των θυμάτων σε περιπτώσεις παραβίασης του ανταγωνισμού ή Δεν θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας μόνο τη συλλογική προσφυγή. Η σημερινή πραγματική πρόκληση αφορά τις ατομικές προσφυγές που ζητούν αποζημίωση περισσότερο και λιγότερο τις συλλογικές. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που χρειάζονται νομοθεσία. Αλλά όχι για τη συλλογική προσφυγή. Εγώ σας ομιλώ τώρα για την ιδιωτική επιβολή ε, του οργανισμού και την αποζημίωση ε, των θυμάτων με ατομική ή ε, συλλογική δράση. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία. Σας ανέφερα προηγουμένως ορισμένα, θα ήθελα επιμείνω σε ένα. Δημοσίευση και αποκάλυψη της ενημέρωσης που έχουμε. σε περίπτωση διερεύνησης των ε, περιπτώσεων στρέπλου στον ανταγωνισμό. Το ε, πρόγραμμα αυτό επιτρέπει να βρούμε τα καρτέλ. Έρχονται σε εμά εταιρείες εμπιστευτικά και μας δίνουν στοιχεία και έγγραφα και στοιχειοδοτούν και αποδεικνύουν την ύπαρξη καρτέλ. Εάν εμείς αποφασίσουμε ότι αυτά τα εμπιστευτικά στοιχεία μπορούν να δημοσιευθούν για οποιονδήποτε ε, ζημιοθέντα που θέλει να κάνει κάποια δράση, χαθήκαμε. Δεν πρόκειται να ξανάρθει ποτέ κανείς. Πρέπει να τους προστατεύουμε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται σε μας. Υπάρχει μια απόφαση ε, δικαστηρίου για μια γερμανική υπόθεση που λέει ότι χρειάζεται δημοθεσία η αρχή υπάρχει και λέει το δικαστήριο το γνωρίζουμε ότι υπάρχει αρχή που προστατεύει αυτές τις εταιρείες αλλά δεν υπάρχει νομοθεσία και το δικαστήριο μας ζητάει να νομοθετήσουμε για την επίκη ε, μεταχείριση ε, αυτών που προσφεύγουν σε μας για να μας καταγγείλουν μια περίπτωση παραβίασης ε, της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Είτε εκ των υστέρων είτε εκ των προτέρων. Λοιπόν, αυτή η νομοθεσία χρειάζεται. Γι' αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουμε για του κανόνε για τι συλλογικέ προσφυγέ τέλη του έτου ή αρχέ επομένου πριν προχωρήσουμε σε νομοθετικά βήματα. Πάντω, σας παρακαλώ ξεχάστε την παλιά πρόταση ή τις παλιές προτάσει που δεν ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2009 εναλλακτική επίλυση διαφορών, το ADR. Συμφωνώ ότι είναι πολύ καλή τεχνική, αλλά με τις ε, περιορισμένες νομικές μου γνώσεις, σε κάποια συντάγματα που γνωρίζω καλύτερα από κάποια άλλα στην Ευρώπη, ουδής μπορεί να πει σε έναν πολίτη, σε μια εταιρεία, ότι δεν δικαιούσε να προσφύγει στα δικαστήρια για να δικαιωθείς. Υπάρχουν τρόποι και μέσα να αποφευθούν περίπλοκες διαδικασίες, καθυστερήσεις, να διακανονιστεί μια υπόθεση πριν το δικαστήριο. Αλλά ε, από το δικό μου νομικό πολιτισμό δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν να απαγορεύει σε ένα πολίτη ή σε μια οντότητα να πάει στα δικαστήρια. Ούτε να του βάλει κανένα φραγμό, εάν το επιθυμεί. Ε, ε, θέλει να προσφύγει και να επικαλεστεί να αξιώσει το δικαίωμα σε αποζημίωση το ενδεχόμενο θύμα. Στην περίπτωση του ADR, της εναρκτικής είπαμε ε, μορφής διευθέτησης, διακανονισμού, ναι, αλλά να μην είναι το μοναδικό μέσο. Μπορεί να είναι καλύτερο, αποτελεσματικότερο, ταχύτερο, αλλά σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Γκογιάνς, ότι δεν μπορεί να βρεθεί διακανονισμό. το ενδεχόμενο ε, θύμα έχει κάθε δικαίωμα να προσφεύγει τη δικαιοσύνη. Αυτή είναι μια αρχή του δικαίου προφανής. Έγινε μια ερώτηση που αφαιρούσε τη Χέγκελ. Δεν είναι θέμα ανταγωνισμού όχι συγγνώμη, την, ε, την Ουγγαρία ε, για τις ε, υποθήκες ή τα δάνεια. Εδώ είναι δύο ζητήματα. Η προστασία του καταναλωτού για να προστατεύονται εκείνοι που έχουν συνάψει στεγαστικά δάνεια και από την άλλη, αν δεν απατώμε, οι ρυθμιστικές αρχές, οι εποπτικές αρχές ή τα χρηματοπιστωτικά συστήματα θα έπρεπε να είχαν προειδοποιήσει για τους τεράστιους κινδύνους για τους πολίτες μιας συγκεκριμένης χώρας όταν έπαιρναν δάνεια με ρήτρα ξένου νομίσματος, ελβετικού φράγκου κλπ. Γιατί ε, το κίνδυνο της ε, συναλλαγματικής ισοτιμίας τον επομίζεται ο καταναλωτής, όχι η τράπεζα. Εσύ παίρνει ένα δάνειο από την τράπεζα, υπογράφεις και σε επιβαρύνει η συναλλαγματική ισοτιμία και η διαφορά στα νομίσματα. Αλλά αυτά είναι θέματα εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα, νομίζω, για την προστασία των καταναλωτών. Δεν είναι θέμα ανταγωνισμού, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής γιατί είσαστε πολύ σαφείς και ήταν πλήρης η αναφορά που μας κάνατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, εύχομαι ότι μαζί με τους συναδέλφους σας Ρέντιν και Ντάλι θα βρείτε ενδιαφέρουσες και ευφυείς λύσεις έτσι ώστε ε, να αποφύγουμε τις τρευλώσεις ε, τις οποίες διαπιστώνουμε στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ναι, θα είναι σίγουρα ευφυείς. Δεν ξέρω αν θα είναι λύσεις, <laughs> αλλά θα είναι σίγουρα ευφυείς, λέει ο κύριος Αλμούνια. Θα δώσω τον λόγο τώρα στον καθηγητή κύριο Ρότς για να απαντήσει ε, στις ερωτήσεις τις οποίες του ετέθησα σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία σημεία. Πρώτα απ' όλα να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Σβάμπ ε, ορισμένες χώρες μέλη έχουν ε, εισαγάγει την ε, διαδικασία συλλογικής προσφυγής. Για λόγους που εξήγησα υπάρχουν και οικονομικά κίνητρα και έλεγχοι στα εθνικά συστήματα. Σε πολλές περιπτώσεις τα εθνικά συστήματα έχουν τελείως διαφορετικούς τεχνικούς ελέγχους για τις συλλογικές προσφυγές. Επίσης διαφέρουν τα οικονομικά κίνητρα αλλά κυρίως ε, δεν θέλουν τα κράτη-μέλη να ε, υπάρξει ενίσχυση της ε, διαδικασίας αυτής προσφυγής και εάν, όπως είπα και προηγουμένως και το εξήγησα, εάν κανείς ενθαρρύνει τα οικονομικά κίνητρα και θα υπάρξουν περισσότερες προσφυγές, αλλά σίγουρα θα είναι υπερβολικά μεγάλος ο αριθμός τους ήδη από αυτό τον πρώτο χρόνο ας πούμε εφαρμογής των συστημάτων ε, βλέπουμε ότι στη Σουηδία, στη, συγγνώμη, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βλέπουμε ότι ε, και υπάρχουν πολύ περισσότερες προσφυγές αλλά και κρατάνε σε μάκρος οι διαδικασίες. Δεν είναι αντίστοιχα ε, τα ε, συστήματα, τα δικαστικά με εξαίρεση ε, την Γερμανία όπου οι διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων είναι σύντομες και αποτελεσματικές. Για μεμονωμένες προσφυγές βέβαια τα χρήματα είναι ακόμα περισσότερα και ο χρόνος ακόμα μακρύτερος. Αλλά εάν θεωρήσει κανείς ότι ισχύει αυτή η κατάσταση στις μεμονωμένες προσφυγές φανταστείτε πόσο περισσότερο περισσότερο περίπλοκο και πόσο περισσότερο ακριβό θα είναι ε, το σύστημα των συλλογικών προσφυγών. Δεύτερο σημείο. Τι είναι παλαιομοδίτικο και τι δεν είναι. Η συλλογική προσφυγή δεν είναι παλαιομοδίτικη, είναι ουσιώδης. Το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστεί. Αυτό που προσπάθησα να πω είναι ότι οι συλλογικέ δράσεις είναι ένα παλιωμοδίτικο μοχλός πίεσης. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα σύγχρονο σύστημα το οποίο θα έχει ένα πρώτο πυλώνα που είναι ε, το διακανονιστικό ε, ε, το εξοδικαστικό, ένα τρίτο πυλώνα που θα είναι τα δικαστήρια και έναν ενδιάμεσο πυλώνα που θα είναι η συλλογική προσφυγή. Δεν θέλουμε το σύστημα να μπλεχτεί στα γρανάζια των δικηγόρων. Ε, βεβαίως μπορεί να υπάρξει ένα νέο σύστημα το οποίο θα βασίζεται στους δύο ακριανούς πυλώνες, θα συρρυκνώσει τον, ε, τον ε, ενδιάμεσο πυλώνα και θα βασιστεί περισσότερο σε ένα σύστημα EDR εναλλακτικών επιλύσεων, εναλλακτικών επιλύσεων διαφορών. Τώρα, όσον αφορά τα κίνητρα, και αυτό είναι το σημείο το οποίο έθιξε η κυρία Γκογιάν, μπορεί κανείς να σχεδιάσει ολοκληρωμένα συστήματα τα οποία ενθαρρύνουν ε, και κάνουν πολύ αποτελεσματικά τα συστήματα ADR αλλά ταυτόχρονα να αντιμετωπίζουν και το άλλο σημείο το οποίο έθιξε η κυρία Γκογιάννη. Δηλαδή, εάν θέλει κανείς να, να χρησιμοποιήσει μόνο τον πρώτο πυλώνα από μόνο του, ε, θα είναι πολύ ακριβό. Εάν θέλει κανείς να χρησιμοποιήσει μόνο τον τρίτο πυλώνα, που είναι τα δικαστήρια, επίσης θα είναι πολύ ακριβό. Και επομένω, το σημαντικό είναι το... Ε, η πονηριά κατά κάποιο τρόπο είναι να μπορέσει κανείς να συνδυάσει αρμονικά τους τρεις πυλώνες και να ξεκινήσει ε, μια, διαδικασία, μια συζήτηση η οποία μπορεί τελικά να φτάσει σε νέες ιδέες όπως ας πούμε είναι ο Δανέζος ε, συνήγορος του καταναλωτή και οπωσδήποτε να ε, υπάρχει μεγαλύτερη κινητροδότηση της εναλλακτική επίλυσης διαφορών του ADR ε, και να κληθούν τα μέλη, τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν ευφιέστερα διαδικασίες οι οποίες έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την προστασία των καταναλωτών. Έχουμε εκτενώς μελετήσει τα συστήματα ADR. Ε, το κάναμε, αυτή τη μελέτη την κάναμε φέτος και στα πρώτους μήνες του επόμενου χρόνου θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα. Το θέμα είναι λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε φιώς τα ήδη υπάρχοντα συστήματα. Τρίτον, Έχω ένα πρόβλημα με την ε, παρούσα στάση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Διότι ξεχωρίζει στην ουσία την δική τους ε, διαδικασία αντιμετώπισης που βασίζεται ε, σε πρόστιμα ε, και σε αποτροπή και αφήνει τελείως στην αγορά το θέμα της ιδιωτικής προσφυγής. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο σύστημα εφαρμογής ε, των ε, πολιτικών, τότε θα πρέπει να δείτε συνολικότερα το δημόσιο και το ιδιωτικό σκέλος. Δηλαδή, να έχουν τη δυνατότητα οι καταναλωτές να κάνουν προσφυγή, αλλά έτσι ώστε αλλά βεβαίως θα πρέπει ε, να ε, υπάρξει και η απαραίτητη εξισορρόπηση της αγοράς. Δηλαδή, εάν ε, πείτε επιβάλλω αυτό το πρόστιμο, δεν είναι βέβαιο ότι η αγορά θα ακολουθήσει και ενδεχομένως να μην υπάρξει και σωστή αποζημίωση στον, προς τους θυγόμενους. Κοιτάξτε, εγώ έγραψα και ένα άρθρο και συγγνώμη που δεν θέλω να κομπάσω, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, ε, έγραψα ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε πρόσφατα και βάσει πινάκων και διαγραμμάτων ε, ακριβώ ακριβώς καταδεικνύεται αυτό που μόλις είπα. Δηλαδή θα πρέπει η πολιτική να μην βασίζεται μονάχα στην αποτροπή και στα πρόστιμα, αλλά και σε άλλα κίνητρα τα οποία είναι πιο σύγχρονα και πιο αποτελεσματικά. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη ε, προσέγγιση που δεν θα βασίζεται ούτε μόνο στα ε, όργανα, ούτε μόνο στα δικαστήρια, ούτε μόνο στο νόμο, ούτε μόνο στα δικαστήρια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Γογιάννης. Ευχαριστώ πολύ. Ένα γενικό θέμα άκουσα σήμερα το πρωί το γεγονός ότι οι συλλογικές προσφυγές αυξάνουν τις διαφορές. Αυτό είναι λάθος προοπτική, λάθος οπτική γωνία. Δηλαδή βασίζεστε στο γεγονός ότι τα μεμονωμένα θύματα δεν προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Μα αυτή δεν είναι δικαιοσύνη. Γιατί στην ουσία ένα σωστό σύστημα μειώνει τις διαφορές διότι ομαδοποιούνται οι διαφορές και έχετε ένα δικαστήριο το οποίο χειρίζεται ε, πολλές διαφορές. Δηλαδή έχουμε έναν εμπειρογνώμονα αντί για εκατοντάδες. Στην περίπτωση του διαμεσολαβητή στη Γαλλία ε, αφορά 500 με 2.000 θύματα. Και εάν είχατε τόσες υποθέσεις τότε πολλαπλασιάζεται το δικαστικό σκέλος επί 500 ή επί 2.000. Το ίδιο αφορά και την ε, Ουγγαρία. Βέβαια, όλοι βασιζόμαστε γεγονό ότι δεν θα προσφύγουν όλοι στη δικαιοσύνη, αλλά αν θέλουμε ένα δίκαιο σύστημα, τότε θα πρέπει να τύχουν αποζημίωση όλα τα θύματα. Και αν υπάρχει ένα συλλογικό σύστημα, τότε γίνεται και πιο αποδοτικό. Το δεύτερο είναι το πορτογαλικό σύστημα. Θα ήθελα να υποθεί ότι το πορτογαλικό σύστημα είναι από τα καλύτερα, διότι είναι ένα πολύ δημιουργικό σύστημα και λειτουργεί πολύ καλά. Δεν οδήγησε σε καμία πτώχευση επιχείρησης, ισχύει εδώ και αρκετές δεκαετίες και ίσως ανέκυψαν 20 υποθέσεις. Και τα δικαστήρια ήταν πολύ δημιουργικά. Ο κύριος Βάμπ μας είπε τι θα γίνει όταν υπάρχουν μικρές, μικρή ζημία. Στην Πορτογαλία έχουμε την υπόθεση Telecom, όπου για μία περίοδο χρεώθηκαν διαφορετικά οι λογαριασμοί. Είναι πολύ δύσκολο για τον καταναλωτή να πει τη συγκεκριμένη στιγμή υπερχρεώθηκα. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι όλοι οι πελάτες αυτής της εταιρείας θα είχαν ε, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο τους χωρίς να πληρώσουν για ένα χι χρονικό διάστημα. Αυτό είναι πολύ δημιουργικό. Και γενικότερα πιστεύω ότι εάν υπάρχει κάποια δυσκολία ποσοστοποίησης ε, της ζημίας των ε, θυμάτων, τότε θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική αποζημίωση, ένα συνολικό σχήμα και αυτό δεν πρέπει να μεταφερθεί στον κρατικό προϋπολογισμό γιατί τότε ίσως υπάρχει ο κίνδυνος να βοηθήσουμε τις ε, τράπεζες οι οποίες αντιμετωπίζουν κάποια δυσχέρεια. Θα μπορούσε να μπει σε ένα ταμείο και αυτό το ταμείο μετά θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει τις συλλογικές προσφυγές για το μέλλον. Αυτό είναι ένα εναλλακτικό σύστημα σε σχέση με την υπόθεση στην Ουγγαρία δεν είναι υπόθεση ανταγωνισμού, αλλά πρόκειται για συλλογική προσφυγή που αναγνωρίζουμε που δεν αφορά ένα σύστημα συλλογικών αποζημιώσεων και συμβαδίζει με τα δικά μας αιτήματα. Θα πρέπει αυτά τα θύματα συλλογικά να μπορέσουν να προσφύγουν στο δικαστήριο. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε για να απαντήσετε στον καθηγητή και να ε, φτάσετε σε ορισμένα συμπεράσματα. Ευχαριστούμε κύριε Γκοζές. Ευχαριστώ κύριε Γκοζές. Μία σύντομη απάντηση και μόνο. Ως προσθέση του καθηγητού Χότζες ως προς αυτά που προείπε για τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Ε, μιλάμε για τρόπο ανάγνωσης των ε, ευρωπαϊκών συνθήκων. Πώς ορίζουμε τον ανταγωνισμό. Είπα στην αρχή ότι θα πρέπει να βρούμε ένα σύνδεσμο μεταξύ δημόσιας ε, συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού και πώς ορίζουμε τις ιδιωτικές προσφυγές. Θα πρέπει να υπάρχει ένας σύνδεσμος και δεν είναι καθόλου εύκολος να οριστεί. Και πράγματι, όλα τα στοιχεία που λάβαμε σε περιπτώσεις συλλογικών προσφυγών που συσχετίζονται με αυτό το θέμα, δηλαδή πώς ορίζουμε την ιδιωτική και τη δημόσια συμμόρφωση, η εφαρμογή, αφορούν ακαδημαϊκούς, εμπειρογνώμονες, εμπλεκόμενους φορείς και ούτω καθεξής. Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη πρόκληση που υφίσταται, έτσι ώστε να υπάρξει αποζημίωση σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων ανταγωνισμού, έτσι ώστε τα θύματα να αποζημιωθούν. Αυτό όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδυναμώσει τη δημόσια εφαρμογή του ανταγωνισμού, δηλαδή την καταπολέμηση των καρτέλ. Η Κομισιόν μπορεί να λάβει τις πληροφορίες που χρειάζεται για τη δική της έρευνα και στη συνέχεια να εφαρμόσουμε τις πιο συνετές λύσεις και τις πιο αποτελεσματικές βεβαίως, έτσι ώστε να μην επιβάλλουμε κυρώσεις στους παραβιαστές, αλλά να αναχαιτήσουμε αυτούς που έχουν αυτό το δέλερ της παραβίασης. Ε, τα αναχαιτιστικά μέτρα, τα μέτρα αναχέτησης είναι πολύ σημαντικά. Όταν οδηγούμε σε ένα αυτοκινητόδρομο και το όριο είναι 120 χιλιόμετρα την ώρα, τότε τα μέτρα αναχέτησης, τα οδικά μέτρα αναχέτησης είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχουν και άλλα σχήματα αν υπάρχει ατύχημα. Συζήτηση με τις ασφαλιστικές εταιρείες και ούτω καθεξής. Αλλά τα μέτρα αναχέτησης είναι πολύ σημαντικά σε περίπτωση δημόσιας συμμόρφωσης. Τώρα, ως προς το ADR, τα, ενα, τις ανελακτικές επιλύσεις διαφορών. Εγώ είμαι υπέρ. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η θέση εκείνων που είπαν ότι το ADR δεν μπορεί να ειδωθεί από μόνο του. Γιατί αν δεν μπορεί κανείς να προσφύγει στα δικαστήρια, τότε δεν είναι παρά ένα πολύ άδικο μέσον. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε και τους παρεμβαίνων για την πολύ σημαντική τους εισφορά. Νομίζω ότι είμαστε ακόμα πιο φωτισμένοι και όταν θα χρειαστεί θα λάβουμε τις αποφάσεις που δεν θα ορίσω, όπως έκανε η κυρία Λούλινγκ που είπε οι σωστές, οι χριστές αποφάσεις. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω τις ε, ημερομηνίες για την προθεσμία τροπολογιών 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Η πρώτη συζήτηση των τροπολογιών θα γίνει στις 11 Οκτωβρίου, η ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ 17 Οκτωβρίου και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια προβλέπεται για το Δεκέμβριο στο Στρασβούργο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. Ο Ανδρέας Βάμπ είναι ο πρωτοπόρος του πρωινού και του αναθέτουμε όλες τις υποθέσεις. Δεν μπορώ να πω βεβαίω ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση και κατά πόσο πρέπει να προβάλλουμε ε, συλλογικές προσφυγές αντιτρά στην περίπτωσή του. Δεν θα ήθελα να φτάσω τόσο μακριά. Λοιπόν, ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ανδρέας Σφάπ είναι ο εισηγητής και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια. Αγαπητέ Ζαν Πολ, μπορώ να σας διαβεβαιώσω από τώρα ότι η ετήσια έγκριση για την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2010 ε, οχριά ε, μπροστά ε, στο six και άλλα τέτοια ελκυστικά ε, νομοθετήματα. Θα δείτε και το ενδιαφέρον των ε, συναδέλφων. Ευχαριστώ λοιπόν για τα λουλούδια που μου στείλατε, αλλά μαραίνονται γρήγορα. Φέτος είναι τα 40 χρόνια της ετήσιας έκθεσης και ο κύριος Αλμούνια είπε ότι ε, εγκρίνονται αυτά του χρόνου και ε, πολλέ φορέ υπάρχει διαφορά μέχρι και δύο ετών ανάμεσα στην έκθεση του Κοινοβουλίου, που έτσι καλώ δεν είναι δεσμευτική, και τα όσα αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλό είναι λοιπόν να αντιδρούμε γρήγορα. Τρία είναι τα θέματα που πρέπει να αναφέρουμε στην ετήσια έκθεση. Πρώτο, ο έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δεύτερο, το δίκαιο για τα καρτέλ και τον ανταγωνισμό και το τρίτο είναι ο διάλογος για τον ανταγωνισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων επικεντρώνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τραπεζικό σύστημα, πώς να ήταν και διαφορετικά άλλωστε για την περσινή χρονιά. Και εμείς καλωσορίσαμε ρητά ε, τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα ε, ε, θεσπίσει κατευθυντήριε γραμμές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των τραπεζών για να έχουν και οι πολίτες τη βεβαιότητα ε, ότι τα χρήματα που δίνουν τα κράτη στις τράπεζες να επενδύονται σωστά και να υπάρχει και απαραίτητη ρευστότητα, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το δεύτερο Υπάρχει ένα καθεστώς προσωρινό για τις κρατικές ενισχύσεις σε περιπτώσεις κρίσης. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά δεν μπορεί να είναι απεριόριστη η ε, παράταση, ούτε ανεξέλεγκτη. Κάποια στιγμή δηλαδή οι κρατικές ενισχύσεις ε, των ε, κρατών μελών στη διάθεση διαφόρων κλάδων της οικονομίας και των τραπεζών θα πρέπει να τερματίζονται και επίσης να αξιολογούνται. Πιάσανε τόπο. Δεύτερον, το δίκαιο ε, για τα καρτέλ, τα είπαμε προηγουμένως σε σχέση με τις συλλογικέ ε, προσφυγές, δεν θέλω να επαναλάβω και να προσθέσω τίποτα, αλλά σε σχέση με κάτι που είπε προηγουμένως ο καθηγητής Χότσης, ε, το ανέφερε ως τρίπτυχο. Επιβολή από το κράτος της νομοθεσίας ως πρώτο πυλώνα, τον τρίτο πυλώνα τον ε, χαρακτήρισε ως τον πυλώνα της αποζημίωσης, αλλά αυτή τη στιγμή στη μέση λείπει μια κολόνα ε, για τους καταναλωτές, αλλά και για τις επιχειρήσεις που έχουν ζημιωθεί, για να μην υπάρχει γραφειοκρατική διαδικασία, να είναι γρήγορη και να αποζημιώνονται καλά. Αυτό το αναφέρω και στην έκθεσή μου, δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλά είναι αυτά που λέει για την αποτροπή, αλλά θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα και ιδιωτικού διακανονισμού ε, να αναζητήσει η εταιρεία ίδια τους πληγέντες και να τους αποζημιώσει. Αυτό είναι πολύ καλύτερο για τους καταναλωτές, πολύ πιο ελπιδοφόρο και πολλά υποσχόμενο από αυτά που είπε προηγουμένως ο κύριος Αλμούνια να καταλήγουν τελικά στα δικαστήρια οι πολίτες. Σημαντικό αυτό. Άλλο σημαντικό. Προτείνουμε στην έκθεση κάτι για τον κανονισμό 1 του 2003. Να συμπληρωθεί η διατύπωση για το πώς υπολογίζονται τα πρόστιμα με τις ε, νέες βασικές αρχές που θα τα διέπουν, όπως είπε ο Επίτροπος. Θα θέλαμε λοιπόν να αλλάξει ο κανονισμός αυτός, ένα του 2003, για να δούμε αυτό που έγινε και στην οικονομική κρίση όλο και περισσότερες εταιρείες επικαλούνται την αδυναμία πληρωμών. Τους έχει επιβάλει ένα πρόστιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτοί σου λένε inability to pay. Δεν έχει βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος επιβολής προστίμων Αλλιώς οι εταιρείε δεν θα ζητούσαν διακανονισμούς και ε, εφαρμογή της αρχής αδυναμίας πληρωμών. Κάτι άλλο που δεν θέλω τώρα να το αναφέρω στην πολιτική ανταγωνισμού είναι η διεθνή συνεργασία. Ε, πάρα πολύ σημαντική. Γιατί εταιρείε από τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, βλέπουν να τους επιβάλλονται πρόστιμα στην Ευρώπη και από άλλες χώρες και η Κίνα και εγώ που είμαι και από παραμεθόρια περιοχή κοντινή με την Ελβετία χαίρομαι που συμμετέχει και η Ελβετία σε αυτή την προσπάθεια γιατί το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού για τα καρτέλ βρίσκει πολύ περιορισμένη εφαρμογή ε, στην Ελβετία γιατί ε, οι αποφάσεις ε, ερεύνης ε, δεν μπορούν να επιβληθούν με την ίδια ταχύτητα και με την ίδια αποτελεσματικότητα όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι μειονέκτημα ανταγωνισμού ή πλεονέκτημα για εταιρείε που έχουν την έδρα του στην Ελβετία. Για τους επιμέρους κλάδους προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τομέα της ενέργειας και δεδομένης και της ενέργειας 2000 και για να τελειώσω, ο διάλογος για τον ανταγωνισμό δεν είναι ένα θέμα με το οποίο μπορούμε να δρέψουμε τεράστιες δάφνες. Τις επόμενες εβδομάδες ε, θα συνεχιστεί. Έχει γίνει με τον Επίτροπο Ολμούνια. Έχω την τιμή να είμαι στην Task Force για την πολιτική ανταγωνισμού και να ε, προεδρεύω και εσείς συμμετείχατε πέρσι. Ε, είχαμε τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού Επαφές με το Γενικό Διευθυντή Ιταλιάνο. Ε, είναι άψογη η συνεργασία μας. Θα κάνουμε και κάποιες προτάσεις για την ετήσια ε, έκθεση για αλλαγή και επευκαιρία τη της 40ης έκθεσης να επικεντρωθούμε ακριβώς στα πιο σημαντικά ζητήματα και να ενισχύσουμε και τις ανταλλαγές για τη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απευθύνομαι και στη συνάδελφο Ινιτφέλτ που πολύ συχνά αναφέρεται και αυτή σε αυτό. Ε, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είμαστε συνομοθέτες, δεν υπάρχει συναπόφαση ε, τα θέματα δικαίου ανταγωνισμού. Σα είπα τα σημαντικότερα που παίζουν ρόλο στην έκθεσή μου. Περιμένουμε ενδιαφέρον να ακούσω του συναδελφού. Σα ευχαριστώ για την προσοχή και ιδιαίτερα για τη συνεργασία με του σκιώδει ηγητέ μέχρι στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ. Βλέπω ότι υπάρχει μία σκιώδης, η Σοφή Ιντβελτ θα είναι και το πρώτο θύμα. Όποιοι θέλουν να παρεύουν, σας παρακαλώ να εγγραφείτε. Σφίμπερκ στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Θα είμαι ιδιαίτερα σύντομη, διότι με μεγάλη μου λύπη έφτασα πολύ αργά και δεν συμμετείχα στο σεμινάριο σήμερα το πρωί, γιατί για τρεις ώρες ε, ακριβώς επειδή υπάρχει, γίνεται μία διαδήλωση. anyway, ε, επειδή γίνεται μία διαδήλωση ε, στο κέντρο των Βρυξελών, γι' αυτό βρεθήκατε τρεις ώρες. Ναι, είναι πολλές, ε, δυστυχώς, είναι πολλές συμφορήσεις κυκλοφορία σήμερα. Ε, εν πάση περιπτώσει, εγκρίναμε την έκθεση ΣΦΑΜ, εξαιρετική ήταν η έκθεση και τα δύο τελευταία χρόνια συνεργαζόμαστε ως εισηγητές και, εισηγητής και σκιώδης εναλλακτικά και υπάρχει μεγάλος ε, βαθμός συμφωνίας στα περισσότερα ζητήματα. Εάν λοιπόν υποβάλουμε τροπολογίες θα γίνουν πολύ μικρές προσθήκες και όχι αλλαγές επί της ουσίας. Ως προς το τελευταίο θέμα που θίξατε για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είμαστε συνομοθέτες, παράλληλα όμως, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση οριμάζει, υπάρχει πολιτική λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του θέματος ε, μέσα στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας. Αυτό θα βοηθούσε όλους. Δεν είναι κάτι το ρίζοσπαστικό. Είναι μία επεξεργασία ή τυποποίηση των ανταλλαγών απόψεων που είχαμε με τον Επίτροπο Αλμούνια μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει feedback στις ετήσιες εκθέσεις μας. Δηλαδή θα, μα θα μας δώσει την δυνατότητα να έχουμε μια πραγματική ανταλλαγή απόψεων και απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί της ουσίας. Η κυρία Σουίνμπερν. Ε, κύριε Γκοζές, ε, ο Σκιώδης έρχεται από την ε, διάσκεψη των Προέδρων. Αν μπορούμε να καθυστερήσουμε λίγο, ακόμα καλύτερα. Εντάξει. Η Ελίζα. Ευχαριστώ κύριε Γκοζές. Παραμβαίνω εξ ονόματος των σκιωδών από τους σοσιαλιστές, αλλά θα ήθελα να πω και κάτι προσωπικό. Ο Πίτερ Σκίνερ είναι σκιώδης, δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα εδώ. Ζήτα συγγνώμη και την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι είναι ευπρόσδεκτη η εργασία του κυρίου Σβάμπ. Προσβλέπει στη συνεργασία μαζί σας και θα ήθελε να τονίσει δύο σημεία που πρέπει να εξεταστούν. Το ένα το προαναφέρατε. Θα πρέπει να εποπτεύουμε τα μέσα κρατικών ενισχύσεων στον τραπεζικό τομέα. Χρειάζονται νέοι κανόνες ε, για να ισχύσουν στον τομέα των χρηματοπιστωτικών ρυθμίσεων και χαιρόμαστε διότι η Επιτροπή ασχολείται με αυτό το θέμα με βάση τις, ε, ε, των νέων υποθέσεων και της νέας νομοθεσίας, των νέων υποθέσεων μάλλον. Το δεύτερο θέμα που έθιξε ο Πίτερ Σκίνερ είναι ένα πρόγραμμα μέτρων και ιδιαίτερα μέτρων επικούς εφαρμογής. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα διαχειριστούμε το θέμα των επιχειρήσεων σε περιπτώσεις, σε υποθέσεις αντιτράστ. Ως προς το θέμα της επίκους μεταχείρισης, αυτό βοηθά ιδιαίτερα τους κοινοποιητές της λειτουργιών και θεωρεί ο Πίτερ Σκίνερ ότι αυτό θα μπορούσε να ενταχθεί στους κανονισμούς και στην όλη διαχείριση από τις γενικές διευθύνσεις προσβλέπει στη στενή συνεργασία. Τώρα εγώ προσωπικά θα ήθελα να τονίσω, μάλλον να παρεκτείνω κάπως το θέμα στον τραπεζικό τομέα, γιατί νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε αυτό τον εναρμονισμένο έλεγχο των, ε, του κρατισμού στις τράπεζες, εάν δεν ενισχύσουμε το διασυνοριακό σύστημα λειτουργίας των τραπεζών και των ελλείψεων που παρουσιάζει. Γι' αυτό περιμένουμε ένα κείμενο. Θα πρέπει να δοθεί μια όθηση, να υπάρχει πολιτική θέληση, έτσι ώστε οι τράπεζες που υπολείπονται σε μέτρα να έχουν, να έχουν αυτή την συνεχή διασύνδεση με τους κρατικούς φορείς, με το κράτος. Γι' αυτό θα θέλαμε η Επιτροπή να προβλέψει κάτι και σε αυτό το τομέα, να νομοθετήσει δηλαδή. Ως προς τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, μας απασχολούν ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Εδώ δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Και Δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα να ζητήσουμε να υπάρξουν τέτοιοι οργανισμοί, ευρωπαϊκοί οργανισμοί πιστοληπτικής ικανότητας. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η άποψη των συναδέλφων. Δεν θα έπρεπε η Κομισιόν να κάνει μία έρευνα και σε αυτή την αγορά που αποκτά άλλο ένα και μεγαλύτερη δύναμη, όπου υπάρχει μαζικός έλεγχος της αγοράς από τρεις επιχειρήσεις, από τρεις οίκους στην ουσία. Αυτό το θέμα θα ήθελα να το εξετάσετε ενδεχομένως, διότι δεν μπορούμε πλέον να το αγνοούμε μέσα στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης ανταγωνισμού. Ο κύριος Λάμπερκ έφτασε, είναι σκιώδης και έχει το λόγο. Δεν ξέρω αν το επιθυμεί πραγματικά. Γιατί ίσως επαναλαμβάνονται πράγματα στο δινικές. Μετά από δύο ε, χρόνια σε αυτή την Επιτροπή έχω κάπως κουραστεί και χειροτερεύουν τα πράγματα με την ηλικία. Δηλαδή τι θες να μου πεις να μην ξαναεκλεγώ. Ε, λοιπόν, αναρωτιέμαι γιατί κάνουμε όλη αυτή τη ε, διαδικασία και θα επαναλάβω αυτά που είπε η Ελίζα πριν από λίγο. Βεβαίως, αντιμετωπίζουμε μια χρηματοπιστωτική βιομηχανία, κυρίως δε τραπεζική βιομηχανία, η οποία ε, δεν μπορεί να παράξει πέρα τις και γι' αυτό εγώ θέλω να θίξω δύο θέματα. Πρώτον, αυτό το ιδιαίτερο πρόγραμμα για την στήριξη των τραπεζών θα πρέπει να διευρυνθεί και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και το, την έκθεση έτσι ώστε ε, να ενισχυθεί από πλευρά τη Επιτροπή η αιρεσιμότητα αυτή τη διαδικασία. Ε, θα πρέπει να πιέσουμε και τις ε, τράπεζες ε, έτσι ώστε να, να επανέλθουν στην αρχική τους πορεία και να αρχίσουν να δανειοδοτούν την πραγματική οικονομία. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμα δυνατότητα βελτίωσης από πλευράς της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνιστικότητας. Δεύτερον, παρά το γεγονός ότι πολύ συχνά το έχουμε αναφέρει ε, η βοήθεια ε, που δίνει η Κεντρική Τράπεζα ε, στις τράπεζες όσον αφορά την ρευστότητά τους, η οποία είναι πρόσκαιρη, μπορεί να δώσει κάποια σταθερότητα στο χρηματοπιστωτικό κλάδο, όμως πιστεύουμε ότι μπορεί να οδηγήσει σε στρέβλωση της αγοράς, σε στρεβλωτικά φαινόμενα. Ακόμα και αν ε, πούμε ότι βραχυπρόθεσμα δεν θα σταματήσουν ή δεν πρέπει να σταματήσουν αυτές οι κινήσεις της Κεντρικής Τράπεζας, παρόλα αυτά θα πρέπει να διαπιστώσουμε νομίζω ότι στρεβλώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την αγορά ε, γιατί ε, κάνει κάποιες παραχωρήσεις ε, προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία ε, χρειάζονται βοήθεια άρα δεν είχαν χρηστή διαχείριση και στην ουσία στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό απέναντι στα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία είχαν χρηστή διαχείριση και δεν χρειάζονται τη βοήθεια αυτή. Ξέρω φλαμανδικές τράπεζες ε, οι οποίες έχουν λειτουργήσει πολύ σωστά και οι οποίες ε, ποτέ δεν ζήτησαν ενίσχυση της ρευτότητάς τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική ε, Τράπεζα γιατί πάντα είχαν πολύ χρηστή διαχείριση. Αλλά εάν ε, δουν ότι ε, στρεβλώνουν το ανταγωνισμό και ότι βρίσκονται σε μειονεκτικό ε, βαθμό ή κατάσταση γιατί δεν προσφεύγουν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα η οποία να τους δώσει δωρεάν στήριξη της ρευστότητας τότε πραγματικά είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι αποδεκτή. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να ξεπεράσουμε τα προβλήματα αυτά και να αντιμετωπίσουμε λύσουμε τα ζητήματα αυτά και με την Κεντρική Τράπεζα και με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όλων των χωρών γενικότερα. Ένα τρίτο σημείο. Ε, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την ε, Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ε, να δει κατά πόσον στη διατραπεζική αγορά υπάρχει χειραγώγηση των στοιχείων. Δηλαδή είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα οποία βιώνουμε τώρα δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας χειραγώγησης και κάποιας τροποποίησης, αλλίωσης των στοιχείων στην διατραπεζική αγορά. Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να να το μελετήσει λίγο. Ε, θα υποβληθούν κάποιες ε, τροπολογίες οι οποίες είναι αντίστοιχες ε, με τροπολογίες που έχουν κατατεθεί προηγούμενα έτη. Βεβαίως η ενέργεια θα πρέπει να καταστεί απολύτως σαφώς, σαφές ότι θέλουμε διαφάνεια ε, εμείς και θέλουμε βεβαίως και να μην υπάρξουν μονοπωλιακές καταστάσεις στο Βέλγιο. Εμείς έχουμε ε, μονάχα έναν κεντρικό operator στο Βέλγιο και αυτό δεν το θέλουμε. Ο Γκιούναρ δεν είναι εδώ, αλλά είναι σαφές ότι ε, χρειαζόμαστε ανταγωνιστική αγορά και η ενέργεια είναι ένας κλάδος, ένας τομέας, στον οποίο πολλά πρέπει και μπορεί να γίνουν θα πρέπει να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην ενέργεια. Ε, επίσης και ο τομέας των τροφίμων. Εκεί βλέπουμε μεγάλους ε, operators ε, οι οποίοι λειτουργούν στα πλαίσια της αγοράς λιανικής και που δεν βοηθούν την διαφάνεια ε, και, την, ε, τον ανταγωνισμό στην αγορά. Βλέπουμε ότι κάποιοι μικρότεροι παίκτες στριμώχνονται υπερβολικά από αυτούς τους μεγάλους ε, και τελικά ο ίδιος ο καταναλωτής ε, πιέζεται πάρα πολύ όπως πιέζονται όπως είπα και προηγουμένως οι μικροί παίχτες σε σχέση με τους μεγάλους. Θα πρέπει να έχουμε πιο ανθεκτική οικονομία και γι' αυτό θα πρέπει να επιτείνουμε τις προσπάθειές μας. Ε, έχει υποθεί κάτι που μου άρεσε παλιότερα ότι ε, θα κάνουμε πράγματα χωρίς να τα ανακοινώσουμε και είπα τι ωραία, θα είναι μια ωραία έκπληξη, αλλά αυτό έγινε πριν από δύο χρόνια και εγώ ακόμα περιμένω την έκπληξη. Μακάρι θα ήταν πολύ ευχάριστο να δούμε την έκπληξη αυτή. Θα υποβάλουμε λοιπόν τροπολογίες κατά αυτή την ε, έννοια, αλλά ειλικρινά ε, κύριοι συνάδελφοι δεν ξέρω κατά πόσον χρησιμεύει σε κάτι όλη αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Φιλίπ. Ο κύριος Επίνγκ. Uh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω να συγχαρώ τον κύριο Σβάμπ για την εργασία του. Υποστηρίζω τα περισσότερα στοιχεία που έχει εντάξει στην έκθεσή του και θα υποβάλω και ορισμένε πρωτοβουλίε. Θα περιοριστώ σε δύο σχόλια. Σε ε, ένα θετικό στοιχείο στην 40η αυτή έκθεση και ένα όχι τόσο ευνοϊκό σχόλιο όλοι ως προσκρατικές ενισχύσεις. Όταν είδα την πανηγυρική σας έκδοση θυμήθηκα ότι η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων ε, και εμπορευμάτων καθώς κεφαλαίων ήταν μια βασική σας πολιτική. Αυτό προωθεί και την ανταγωνιστικότητα, τον ανταγωνισμό εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποίησε όλο ένα και περισσότερο το μηχανισμό αυτό των οικονομικών αναλύσεων και ελπίζω το ίδιο να κάνει και για το μέλλον. Όταν πρόσφατα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έθιξε, μάλλον έκρουσε τον κόδωνα κινδύνου για τις ευρωπαϊκές τράπεζες ένα μήνα πριν, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μας έδωσαν, μας προέβαλαν εγγύσεις δύο μέρες πριν. Σύμφωνα με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι ευρωπαϊκές τράπεζες κεφαλαιοποιούνται πολύ καλύτερα από δύο χρόνια πριν. Όμως σήμερα ο κύριος Αλμούνια τόνισε ότι θα πρέπει να επανακεφαλαιοποιηθούν πολλές τράπεζες που δεν τα κατάφεραν στο τεστ δοκιμών τον Ιούλιο. Πρόκειται για εννέα τράπεζες και αυτό σε σχέση με το 2008-2009, έτσι ώστε οι τράπεζες μπορούν να ενισχύσουν, τα κράτη να μπορούν να ενισχύσουν τις τράπεζές τους μέσα στο 2011. Επίσης υπάρχουν ε, προσωρινά μέτρα τα οποία μπορεί να μην είναι καθόλου προσωρινά μακροχρόνια. Επίσης, το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις στο δινεκές και προσωρινά μέτρα. Σήμερα μιλάμε για μια νέα παράταση του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων, το οποίο υποτίθεται θα ήταν προσωρινό. Άρα βλέπετε ότι η λέξη προσωρινό όλο και επαναλαμβάνεται και ισχύει στο δινεκές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, καμιά φορά ε, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Ο κύριος Φάπ έχει το λόγο για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στα γαλλικά. Ε, επειδή είμαστε μεταξύ μας, ε, να τα πω αγγλικά. Ε, Φιλίπ, ε, δεν είναι ότι το θέμα είναι βαρετό, αλλά κάθε χρόνο ε, όλοι οι συνάδελφοι φορτώνουν την έκθεση με το τι πρέπει να γίνει. Και αυτό είναι κίνητρο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το στείλει το κείμενο κατευθείαν στο κάλαθο των χρήστων. Εμείς φταίμε που δεν είναι σημαντικές οι εκθέσεις αυτές. Μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα αν θέλουμε και προσωπικά πιστεύω ότι γίνεται. Πρέπει να σας πω ότι εκπλήσωμε. Ο κύριος Αλμούνια θεωρεί ότι είναι μεγάλο πρόβλημα οι ε, προτάσεις του κυρίου Χότζες, αλλά κανείς δεν έκανε, έβγαλε κύχ Τι λέει ο κύριος Χότζες, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει τους καταναλωτές να αποζημιώνεται θα πρέπει ε, πριν επιβάλλει το, το πρόστιμο να ορίσει ένα μηχανισμό ADR. Ο Αλμούνια διαφωνεί ε, και κανείς δεν βγάζει λέξη. Το άλλο με τις κρατικές ενισχύσεις δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά. Εμένα με ενδιαφέρει γιατί είναι προβληματική τομή. Μην ανησυχείς, δεν τους υποτιμώ. Απλώς να λέμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα στα α, β, γ, δ δεν βοηθάει. αν βάλουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις τρευλώσεις της αγοράς με τις βοήθειες που παρέχει σε μεγάλες τράπεζες, εντάξει, αλλά θα ζητήσω από τους συντονιστές να κάνουμε έκθεση ιδέα πρωτοβουλίας για να διευρυνθεί η προσπάθεια αυτή και να εμβαθυνθεί. Όχι να το θίγουμε απλώς και περνάμε στην επόμενη χρονιά. Αυτό ισχύει επίσης και για τα διατραπεζικά επιτόκια, αλλά δεν έχει νόημα να τα βάλουμε παρόδο ε, και να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη μετά σε αυτή την έκθεση. συμφωνώ ε, και χαίρομαι για αυτά που λέτε και τα επίμαχα, αλλά θέλω να τονίσω ότι ε, είναι σημαντικό και το στοιχείο των καρτέλ και η καταπολέμηση των τραστ στην έκθεση και πριν την οριστικοποιήσουμε θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως χρειάζεται μια συζήτηση για το σύστημα ε, των συλλογικών προσφυγών. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα καρτέλ. Δηλαδή, όταν έχει διαπιστωθεί ένα καρτέλ, να αποζημιώνονται πρώτα οι πληγέντες και μετά να καταλήγουν για το πρόστιμο. Βέβαια, η Κομισιόν σου λέει ότι αυτό είναι για αποτροπή το πρόστιμο, δεν είναι για αποζημίωση των θυμάτων. Και είναι γεγονό. Στο τέλο μπορεί να μην έχουμε λόγο δικαστικό ή νομικό, αλλά πολιτικό πώ και είναι σημαντικό αυτό. Για όλα τα υπόλοιπα, σας είπα, είμαι πρόθυμος να συνεργαστούμε και σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Και αυτά που είπε η Σοφή για μεγαλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, είπες για τη διοργανική συμφωνία. Εγώ πιστεύω ότι απέχουμε πόρο ακόμα. Το πρόβλημα δεν είναι το κοινοβούλιο, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε πιο συγκεκριμένες προτάσεις, τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να αναμένουμε γιατί κανονικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενημερώνει αλλά χάνεται κάπου ε, στο χωνευτήρι των σημαντικών εγγράφων του Κοινοβουλίου. Είναι καλή συζήτηση, σημαντική. Εγώ δεν είμαι κουρασμένο, Φίλιππ, δεν έχω κουραστεί. Ε, σε ενθαρρύνω να με βοηθήσει κι εσύ αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Σιγητά. Θέλει κανείς να απαντήσει επί προσωπικού. Όχι, συμφωνεί ο Φιλίπ, θαυμάσια. Τελειώσαμε νωρίτερα. Η επόμενη έκθεση έχει προβλεφθεί για τις 11.30 ε, και ο εισηγητής απουσιάζει, δεν μπορώ να προτάξω το θέμα του. Η ψηφοφορία είναι στις 12 παρατέταρτο. Λοιπόν, διακοπή της συνεδρίας μέχρι τις 11.30. Τι να κάνουμε. Α, ξέχασα, ξέχασα, συγγνώμη να σας πω. Ε, προθεσμία για τι τροπολογίε για την έκθεση ΣΒΑΠ 30 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα, συζήτηση για τι τροπολογίε 17 Οκτωβρίου, η ψηφοφορία στην Οικονομική Επιτροπή 22 Νοεμβρίου και στην Ολομέλεια στη δεύτερη του Δεκεμβρίου. Διακοπή της συνεδρίας μέχρι τις 11.30. Σα ευχαριστώ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ.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 Ευχαριστώ. Συνεχίζεται τη συνεδρία, συζητώ συγγνώμη, αλλά νόμιζα ότι δεν θα προείδρευα εγώ πια και θα ερχόταν η Άστρετ στις 11.30. Ε, είχα χαλαρώσει λίγο, αλλά <laughs> ξεχάστηκα. Λοιπόν, ξέρουμε ότι έχουμε ψηφοφορίες παρατέταρτο, αλλά προηγουμένως μικρή συζήτηση για την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Διάσταση του Αθλητισμού. Ο συνάδελφος Μπούρχαρτ Μπάλτς είναι στον Ουάσιγκτον σε αποστολή και θα μας τα πει η κυρία Ισαΐα η οποία ε, είναι και ειδικό επαΐων για αυτά τα θέματα και θα μας ε, παρουσιάσει την έκθεση του κυρίου Μπάλτς στα αγγλικά. Ο κύριος Βάλς, λοιπόν πρώτα απ' όλα ήθελε να σας ευχαριστήσει και να ευχαριστήσει και όλους τους οι εισηγητέ και όλους αυτούς οι οποίοι υπέβαλαν τροπολογίες ε, στην ε, γνωμοδότησή του δίνοντάς της ε, μεγαλύτερο εύρος και βάθος. Έχουμε κάποιες προφορικές τροπολογίες, τέσσερις προφορικές τροπολογίες, και επίσης στις 8 και 21, 20 ε, μάλλον έχουμε μια απλώς καλύτερη διατύπωση αλλά τα, η ουσία ε, παραμένει η ίδια και επομένως μπορούμε να δεχτούμε τις τροπολογίες αυτές. Τροπολογίες 9 και 17 ε, εκεί γνωστοποιείται ότι κάποιες ε, χώρες έχουν μονοπόλιο στα τυχερά παιχνίδια ε, και επομένως θα πρέπει όπως αναφέρεται και στο, στην τροπολογία 9 δεν αρνούμεθα τα, το δικαίωμα στις, στην αποζημίωση όσον αφορά in a little bit different way. So those issues ε, ε, έχουν δικαίωμα λοιπόν να αποζημιώνονται από τα γραφεία στοιχημάτων ε, οι, όλοι οι αθλητικοί φορείς και οι διοργανωτές αθλητικών οργανώσεων. Δεχόμαστε τις τροπολογίες αυτές γενικώ. Ευχαριστούμε πολύ. Σχόλια ενδεχομένως. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Όχι. Τι να κάνουμε, να περιμένουμε να έρθει ακριβώς η ώρα. Όχι. Να ψηφίσουμε λοιπόν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 κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 8 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2α, τροπολογία, ε, επί της τροπολογίας 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 18, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 19, υπέρ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Πάω πολύ γρήγορα. Έκανα λάθος. Επανερχόμεθα λοιπόν. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην παράγραφο 3. Είναι η δεύτερη σελίδα που μου διέφυγε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, παράγραφος 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 11, τροπολογία 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 συμβατή με τη 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 επίσης συμβατή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και μετά να ψηφίσουμε on block για όλες τις υπόλοιπες τροπολογίες. Συμφωνείτε όλοι. Εντάξει λοιπόν, από την παράγραφο 7 μέχρι και την τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Άψογοι είμαστε. Ψηφίζουμε τώρα στο τροποποιημένο κείμενο, για το τροποποιημένο κείμενο υπέρ κατά αποχές δεν υπάρχει καμία αποχή, επομένως εγκρίνεται ομόφωνα το κείμενο αυτό και συγχαιρόμαστε τον κύριο Μπουκχαρτ Μπάλτς. Τώρα, ψηφοφορία επί της εκθέσεως Κάζα σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ. Εδώ θα προσπαθήσω να βρω τις σελίδες μία προς μία για να μην πηδήξω πάλι τροπολογίες. Ε, αρχικό κείμενο για τον υπότιτλο 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι άλλες τροπολογίες. Τροπολογία 12 υπέρ. Ναι, με προφορική τροπολογία του εισηγητού, την οποία γνωρίζετε ήδη, υπέρ, κατά αποχές, Ναι. Δεν βλέπω πώς ψηφίζει το ΕΛΚΑ. Δεν έχει σημασία. 12, 13, συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά απορρίπτεται. Παράγραφος 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική C υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά κατά κατά Α, εντάξει, εγκρίνεται. Όλοι ήταν υπέρ. Συμβεβαστική τροπολογία D, λατινικό, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, Τροπολογία 16, γνωμοδότηση Τσίμκο, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10, ε, γνωμοδότηση των μεταφορών, υπέρ κατά εγκρίνεται. Α, απορρίπτεται. Εντάξει, απορρίπτεται. Η τροπολογία 10 απορρίπτεται. 27, υπέρ... Α, συγγνώμη, 24 λέει ο πρόεδρος. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να επανεκλεγώ και στην επόμενη θητεία για να μπορέσω να τα κάνω καλά όλα αυτά. 24 λοιπόν υπέρ κατά από. Οι φιλελεύθεροι υπερψηφίζουν. Λοιπόν, να ελέγξουμε. Θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Να βρω και εγώ την κάρτα ψηφοφορίας μου. Ψηφίζουμε επί της τροπολογίας 24, έτσι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 18 υπέρ 13 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 25 συμβατή με την 24. Πώς είπατε. Νομίζω ότι επί της τροπολογίας 4 ε, είπατε ότι εγκρίνεται η τροπολογία. Ναι, ναι, αρέ μου, θα ελέγξουμε, λέει ο Πρόεδρος. Ε, εγώ σας σέβομαι, αλίμονο. Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ μια ανοιχτής δημοκρατίας. Θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση επί του 4, αφού λέτε ότι είναι ίδια ε, πλειοψηφία με την τροπολογία 10. Τροπολογία 4, λοιπόν, η γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών ε, και αν καταλάβετε ότι η ταπεινότητά μου έκανε κάποιο λάθος, παρακαλώ να μου το πείτε αμέσως. Πέρας της ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 12 κατά. Εγκρίνεται. Βλέπετε. Διάξτε, είναι οικονομολόγος ο συνάδελφος και νομίζω ότι ε, ε, έτσι όπως έχουν τα πράγματα τώρα δεν πρέπει να τους εμπιστευόμαστε αυτούς τους οικονομολόγους. Λοιπόν, τροπολογία 25 ε, ε, λοιπόν, η αριστερά προσπαθεί να με ε, ενοχλήσει έτσι ώστε να τα χάσω λίγο, αλλά εγώ εκεί 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 27 υπέρ κατά απορρίπτεται, 28 υπέρ κατά απορρίπτεται, 29 με προφορική τροπολογία του εισηγητού υπέρ Θέλετε να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία, ωραία. Υπέρ της ε, προφορικής τροπολογίας. Κατά. Κατά. Ε, ναι, πρέπει να συμφωνήσετε. Η ίδια το ΕΛΚ δεν ξέρει πώς θα ψηφίσει. Το ίδιο γίνεται και στη Γαλλία. Λοιπόν, ποιος είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας. Είμαστε κατά της προφορικής τροπολογίας, λέει ο κ. Καντάου. Ποιο είναι υπέρ τη προφορικής τροπολογίας. Α, δεν θέλετε να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία. Όχι. Ε, είμαστε κατά αυτή της προφορικής τροπολογίας, λέει η κυρία ε, Μπερέσε, ε, πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρέπει να ψηφιστεί αυτή η προφορική τροπολογία. εντάξει, λέει ο πρόεδρος, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ε, ωραία. Υπέρ λοιπόν, χωρίς την προφορική τροπολογία, υπέρ κατά εγκρίνεται. Το, η τροπολογία 20 καταπίπτει, συμβιβασμός ε, υπέρ κατά εγκρίνεται. Παράγραφος 7 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός F λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβιβασμός G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 είναι συμβατή, επομένως ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 επίσης συμβατή υπέρ κατά απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 43 υπέρ κατά εγκρίνεται, 44 υπέρ κατά εγκρίνεται, Συμβιβασ... αρχικός κείμενος, ε, αρχικό κείμενο συγγνώμη, του υποτίτλου 3 υπέρ κατά εγκρίνεται, ε, συμβιβασμός H ε, λατινικό υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 13, ναι. Τροπολογία 13, γνωμοδότηση της ΣΥΜΚΟ υπέρ, κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας 17 υπέρ, 15 κατά, εγκρίνεται. Εγκρίνεται η τροπολογία 13. Τροπολογία 15. Ε, συμβατή με την τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, ε, συμβιβασμός I υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Συμβιβασμός J υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 56 συμβατή και αυτή υπέρ, κατά εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο του υποτίτλου 4 υπέρ κατά εγκρίνεται. Ε, συμβιβασμός K υπέρ κατά εγκρίνεται. Έλεγχος του προϋπολογισμού έχει υποβάλει η Επιτροπή αυτή. Τροπολογία 2. Θέλετε on block. Μπορούμε να ψηφίσουμε από τη 2 μέχρι την 9. Λοιπόν, τροπολογίες. Τροπολογίες από το 2 μέχρι το 6. Τροπολογίες 2 μέχρι 6 υπέρ κατά εγκρίνονται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά απορρίπτεται. 8 και 9 μπλοκ υπέρ κατά εγκρίνονται. 10, 11, 12 μπλοκ υπέρ κατά απορρίπτονται. Συμβιβασμός L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 συμβατή και αυτή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο υπότιτλος 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός M υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ κατά απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 γνωμοδότηση της ΣΥΜΚΟ καταπίπτει, συμβιβασμός N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ναι, όχι. Ωραία, ωραία. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 68. Πέρας της ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 18 ψήφοι υπέρ, 13 ψήφοι κατά, επομένως εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καράσα. Τώρα έχω το νου μου. Συμβιβασμός Α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αρχικό κείμενο ιδεολογική σκέψη B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 8 υπέρ κατά α, εγκρίνονται. Συμβιβασμός Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 επί του νέου ΣΥΑ υπέρ κατά α, απορρίπτεται. Α, κύριε Βαγκόκ, συμφωνείτε, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Αρχικό κείμενο από τις ε, Παύλες 3 μέχρι 9 υπέρ κατά εγκρίνονται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γνωμοδότηση ελέγχου του προϋπολογισμού 0 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και επομένως φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία. Θα γίνει ε, με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία επί του τελικού κειμένου. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν με 30, φο... 30 ε, ψήφους υπέρ και μία ψήφο κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Κάζα, ο οποίος έδειξε τουλάχιστον ότι εκείνος έχει ΦΠΑ, έχει προστιθέμενη αξία τουλάχιστον. Έκθεση Giggold, θα ψηφίσουμε. Ε, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 επί των άρθρων υπέρ. Τροπολογία 4 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Α, θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση, παρακαλώ. Δεν νομίζω ότι έκανα λάθος αυτή τη φορά, αλλά θα το δούμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεν είναι τροπολογία του εισηγητού. 14 ε, ψήφοι υπέρ, 17 κατά, επομένως απορρίπτεται. Τροπολογία 5 του κυρίου Λιέμ Χοάνγκ Νγκόκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 του ιδίου συγγραφέως υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 μαζί με τις άλλες τροπολογίες 9 και 11, 9 και 11 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Μετά τροπολογίες 8 και 10 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε επαλήθευση. Ωραία. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ο, τροπολογίες 8 και 10. Εδώ είναι στρογγυλή η αίθουσα και μπερδεύομαι λίγο. Δεν μπορώ να μετρήσω όλες τις ψήφους και να δω πώς ψηφίζει ο καθένας. Λοιπόν, 28 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά Κοιτάξτε, ε, είδα ότι όλοι όσοι προεδρεύουν σε αυτές τις ε, επιτροπές υπάρχει μία περίπτωση που ο πρόεδρος δεν έχει δει καθόλου καλά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Άλλη φορά δεν θα κοροϊδέψω κανέναν. Λοιπόν, τροπολογία 3, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροποποιημένο κείμενο, ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται, πέρας της ψηφοφορίας. 30 ψήφοι υπέρ, ε, μία ψήφος κατά, καμία ε, αποχή και επί του νομοθετικού ψηφίσματος πάλι διελεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρα της ψηφοφορίας. Α, δεν ψήφισαν όλοι. Τώρα ψηφίσατε. Πέρα της ψηφοφορίας. 27 ψήφοι υπέρ. Μία αποχή. Συγχαίρουμε τον κύριο Γκίγκολτ για την εξαίρετη έκθεσή του. Τελειώσαν οι ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ξαναπάτε τώρα στα μποτιλιαρίσματα. Αλλά έχουμε τώρα την έκθεση του κύριου hans Πέτερ Μάρτιν για την έκδοση κερμάτων ευρώ. Είναι εδώ ο κύριος Μάρτιν. Εδώ είναι. Α, κρύβεστε εκεί πίσω. Κύριε Σιγητά, έχετε δύο εκθέσεις, 7 και 8. Συνδέονται οι δύο κανονισμοί. Κύριε Σβάμπ, μπορείτε να μην μου κρύβετε τον κύριο Μάρτιν να βλέπω τον εισηγητή. Έχει κλέψει την παράσταση έτσι κι αλλιώς σήμερα το πρωί, δεν χρειάζεται και τώρα. Λοιπόν, παρακαλώ κύριε Μάρτιν να μας παρουσιάσετε αν θέλετε και τις δύο εκθέσεις σας, γιατί συνδέονται εκτός αν έχετε αντίρρηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βλέπουμε ότι όταν πρόκειται για το χρήμα δεν είναι τόσο σημαντικό ίσως όσο φαίνεται, γιατί αδειάζει η αίθουσα. Αλλά είναι διοικητικά, θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Γιατί όμως στα χέρια των πολιτών μπορεί να έχουν περισσότερη επίδραση από ό,τι ορισμένα που μας απασχολούν. Είναι δύο κανονισμοί, όπως είπατε, μια νομοθετικού περιεχομένου και μια μη νομοθετικού περιεχομένου για την έκδοση κερμάτων ευρώ. Τα βασικά σημεία είναι ακριβώς και στους καιρούς που ζούμε θα είχε νόημα να τηρήσουμε τις αρχές μας και να πούμε ότι θέλουμε να εξακολουθήσουμε να έχουμε μια ουδέτερη και ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρμόδια για την κυκλοφορία του νομίσματος και ενδεχομένω να έχουμε και ένα χαρακτηριστικό του πληθωρισμού, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ε, τι ενδιαφέρει την έκθεση. Είναι τρία είδη κερμάτων, τα κανονικά κέρματα, τα συλλεκτικά και τα αναμνηστικά και τι θα πρέπει να εκδίδεται σε κάθε κατηγορία. Έχει σημασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει λόγο και σε αυτά τα θέματα, όχι μόνο στον έλεγχο ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι αυτά. Θα ήθελα να επαναλάβω μια ιδέα που κυκλοφορεί σε αρκετές χώρες για το θέμα των ε, χαρτονομισμάτων. Ε, έρχομαι από τι Ηνωμένε Πολιτείε γιατί είχα πάει για μια κηδεία ε, και ξαναμπαίνει το ζήτημα των χαρτονομισμάτων για το 1 ευρώ και τα 2 ευρώ. Γιατί να έχουν στην Αμερική τόσο μικρά χαρτονομίσματα και να μην έχουμε εμεί, Γιατί είναι και μεγάλο το κόστος κοπής νομισμάτων, κερμάτων. τα άλλα θέματα είναι πιο τεχνικά και πιο διευκρινιστικά Και επίση θα πρέπει να δούμε λίγο και τα σχέδια να είναι κοντά στον πολίτη, αυτά που απεικονίζουν τα ευρώ. Θα μπορούσα να φαντάζομαι ένα ισπανικό νόμισμα ευρώ που να έχει σχέση με δημοκρατία ή ε, ένα γερμανικό με τη ε, επανάσταση των αγροτών ε, ή κάτι άλλο αντίστοιχο στην Αυστρία. Δεν το λέω ειρωνικά. Δεν έχει να κάνει ε, με το κεφαλή της χώρας, τον πρόεδρο της χώρας. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα δεν είναι να έχω την κεφαλή του ηγέτη, αλλά κάτι που έχει βοηθήσει και έχει οδηγήσει ε, στην Ευρωπαϊκή Ενωπίωση. Το 1848 ε, ξεκίνησαν ε, ε, στη χώρα μου τέτοιες προσπάθειες ενώ είχε προηγηθεί η Αμερική, οι Ηνωμένε Πολιτείε ως προς την ανεξαρτησία. Επίσης θα πρέπει να προσέξουμε να μην έχουμε ε, σύμβολα επιθετικά που να ακριβώς επιτίθενται σε άλλους λαούς. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα κάποιοι φραγμοί στα μυαλά και δεν ε, είναι πάρα πολύ ανοιχτό το πνεύμα όλων και θέλω να έχει λόγο και το Κοινοβούλιο, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν κατάλαβα αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα συλλεκτικά νομίσματα που ουσιαστικά τα αφήνουμε στην άκρη. Δεν θα πρέπει, λέει, να έχει ε, το ισπανικό άνθος που απεικονίζει, δεν κατάλαβα. Γιατί πρέπει να είναι διαφορετικά τα αναμνηστικά και τα συλλεκτικά για να μην μπορούν να χρησιμοποιούνται ως κανονικά νομίσματα. Μην διαφέρουν τόσο πολύ ώστε να μην μπορούν να κυκλοφορούν. Επειδή είναι 12 και 5 και όχι 12 παρά 5, θα σταματήσω εδώ ε, για να μπορέσουν να μιλήσουν και οι συνάδελφοι, εξή τρει, δηλαδή τέσσερι μαζί με τον πρόεδρο. Αυτή είναι η κατεύθυνση, ελπίζω να συμφωνήσουν και οι συνάδελφοι και αρχές Οκτωβρίου θα σας έχω και την επόμενη έκθεση. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο πρώτα στους κοιόδης ηγητές, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ελπίζω να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον εισηγητή και ότι θα προχωρήσουμε καλά από κοινού και ότι θα φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Η Σοφή δεν έχει τίποτα άλλο να πει. Τα είπε όλα για τον ανταγωνισμό και έκλεισε. Γκίγκολτ ε, δεν είναι εδώ, ούτε ο άλλος συνάδελφος. Κάποιος άλλος που θέλει να... Ο κύριος Γκίγκολτ είναι εδώ, δεν τον βλέπω. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο. Εγώ επειδή αφαιρέθηκα λίγο, θα ήθελα να μου πει ο εισηγητής ποια είναι η θέση του. Μίλησε γι' αυτό για το νόμισμα του ενός ευρώ. Είναι ένα θέμα που έχει ήδη θυγεί και στη Γαλλία. Υπάρχει μία επιτροπή ε, που απαρτίζεται ε, μεταξύ άλλων από το γιο του πρώην Προέδρου του Ζισκάρ Ντεστά έτσι ώστε να εκδοθεί χαρτονόμισμα του ενός ευρώ. Ε, εγώ ήμουν υπέρ αλλά η έκτα αντιτίθεται και δεν άκουσα τη δική σας θέση και ζητώ συγγνώμη. Τι είπατε για την έκδοση χαρτονομίσματος ενός ευρώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Yeah, uh, είναι πάρα πολύ δημοφιλές αυτό το θέμα. Δεν θα έλεγα ότι είναι δημαγωγικό από πλευράς ε, πρακτικής εφαρμογής προσωπικά είμαι υπέρ του τραπεζογραμματίου του ενός ευρώ. Βέβαια θα έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής στα τα χαρτονομίσματα. Αλλά έχει αυξηθεί και το κόστος ε, κοπής ε, κερμάτων. Ας το δοκιμάσουμε να δούμε πώς έχουν οι σχετισμοί και οι πλειοψηφίες στην Επιτροπή μας. Νομίζω αυτό είναι ένα στοιχείο που ζωντανεύει τη συζήτηση όταν συζητάμε με πολλούς πολίτες. Στην έκθεσή μου θα βρείτε τροπολογία σχετική ε, προς την πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την κατεύθυνση αυτή. Υπό κάποιου όρου θα ζητάει να ε, έχουμε χαρτονομίσματα του ενός και των 2 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω ότι θα υποστήριξω αυτή την τροπολογία για πολλούς λόγους. Και για ένα συμβολικό λόγο το χαρτονόμισμα έχει άλλη βαρύτητα από ότι το κέρμα. Έτσι κάνει μεγαλύτερη εντύπωση. Η απόδειξη είναι ότι οι ΗΠΑ έχουν και χαρτονόμισμα ενό δολαρίου. Και για εκείνου που ταξιδεύουν, όταν δίνει πουρμπουάρ σε ευρώ, σε κέρμα, δεν μπορούν να το αλλάξουν. Πρέπει να βρουν κάποιον να το αλλάξει, να του το κάνει χαρτονόμισμα, γιατί δεν μπορούν να το αλλάξουν μετά. Είναι παράδοξο αυτό. Βέβαια δεν αφορά όλου έχουν όλοι μαζί τους δολάρια, ε, ε, μικρά νομίσματα για να δίνεις ε, δολάρια φιλοδόρημα. Θα ήταν καλύτερο να είναι ευρώ αυτά τα μικρά χαρτονομίσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πει τίποτα. Θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που έχουμε αυτή τη συζήτηση με το Κοινοβούλιο. Για πρώτη φορά το Κοινοβούλιο αποφαίνεται σε ένα τέτοιο θέμα για τα μετρητά, τα ευρώ, γιατί δεν υπήρχε νομική βάση μέχρι τώρα. Εντάχει μερικά σχόλια στις παρατηρήσεις του εισηγητή σας ως θεματοφύλακας των συνθήκων θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση νομικής υφής. Η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου για την περίπτωση χαρτονομίσματος του ενός ευρώ θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε ένα ψήφισμα. Δεν μπορούμε να δυσαγάγουμε με βάση τροπολογίας, διότι τα θέμα, τον, το θέμα της έκδοσης χαρτονομισμάτων εξαρτάται αποκλειστικά από την ΕΚΤ. Γι' αυτό είναι αδύνατον να εισαχθεί ένα τέτοιο δεσμευτικό στοιχείο στο κείμενο κάθε αυτό. Από τεχνικής πλευράς θα ήθελα να πω ότι τα νομίσματα του ενός ευρώ είναι αναγκαία αυτή τη στιγμή για την συνολική έκδοση και κοπή αυτών των νομισμάτων γιατί ξέρετε ότι υπάρχει, υπάρχουν κέρδη και στην κοπή. Εν πάση περιπτώσει, το νόμισμα του ενός ευρώ φυσικά φυσικά στοιχείς πολύ περισσότερο. Σε σχέση με τα συλλεκτικά νομίσματα είναι γεγονός ότι δεν γίνεται λόγο στο κείμενο που σας έχει υποβληθεί γιατί αυτό το κείμενο βασίζεται στο προϋπάρχον πλαίσιο. Δεν μπορεί να υπάρχει ρύθμιση για τα συλλεκτικά νομίσματα Θεωρούμε όμως ότι αυτά τα νομίσματα αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένα και δεν θα θέλαμε αυτά τα νομίσματα να συγχέονται με τα κοινά νομίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται στις τρέχουσες συναλλαγές. Με μεγάλη χαρά όμως να το συζητήσουμε με τον εισηγητή και του σκιώδη, καθώς και με τα μέλη της Επιτροπής σας. Ευχαριστούμε την Επιτροπή για αυτή τη νομική υπενθύμηση. Ξέρετε όμως ότι στο Κοινοβούλιο εισαγάγουμε σε κείμενα κάτι σαν ευσεβείς πόθους, χωρίς να έχουμε ε, καμία αυταπάτη σε σχέση με τη νομική υφή του θέματος. Ο εισηγητής θέλει να πει κάτι άλλο. Εν κατακλείδη όχι, φαίνεται πως όχι. Σας ευχαριστώ. Χρονοδιάγραμμα. Η έκθεση θα υποβληθεί στις 24 Οκτωβρίου 2011. Προθεσμία για τροπολογίες 28 Οκτωβρίου. Συζήτηση για τις τροπολογίες 22 Νοεμβρίου. Θα ψηφίσουμε στις 29 Νοεμβρίου στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια θα ψηφιστεί η έκθεση το Φεβρουάριο του 2012. Αυτά και με αυτά τα θέματα σας ευχαριστώ πολύ κύριε εισηγητά και σας εύχομαι κάθε επιτυχία για τη συνέχεια. Υπάρχει τίποτα άλλο στα διάφορα. Από τη δική μου πλευρά δεν υπάρχει τίποτα. Άρα το επόμενο θέμα, πότε θα γίνει η επόμενη μας συνεδρίαση στο Στρασβούργο θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Θα θα πούμε λοιπόν με την πρόεδρο. 8.30. Το... 8,5. 8,5. 8,5. Μέχρι τις 8.30 με συγχωρείτε. Χαίρετε.